Καλημέρα. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίση μας σήμερα το πρωί. Πρώτα απ' όλα βέβαια, θερμό καλωσόρισμα στον Σεβαστιάν Πινιέρα, τον πρόεδρο της Χιλής. Είναι αλήθεια ότι πολύ καιρό δεν είχαμε πρόεδρο της Χιλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, είναι μεγάλη ικανοποίηση για μας να σας έχουμε μαζί σας, εσά και την αντιπροσωπεία σα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αλφρέντο Μορένο και τον πρέσβη της Χιλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Κάρλο Σαχέλη. Είναι ένα πολύ καλό εταίρο της Ευρωπαϊκή Ένωση η Χιλή. Επικυρώσαμε μια συμφωνία που έχει καρποφορήσει και για τις δύο πλευρές. Ενισχύθηκαν οι εμπορικές μας σχέσεις, ο πολιτικός διάλογος αλλά και η συνεργασία. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι η πιο φιλόδοξη από όσε έχει συνυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια τρίτη χώρα. Είναι μία από τι συμφωνίε τέταρτη γενιά, όπω τι ονομάζουμε. Στα πλαίσια τη συμφωνία αυτή, ένα βασικό στοιχείο είναι ο πολιτικό διάλογο. Εμεί ω Ευρωβουλευτέ θέλουμε να υπογραμμίσουμε όλο ιδιαίτερω την διάσταση του διαλόγου αυτού και έχουμε και τον πρόεδρο Κάμπος εδώ που είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τον βουλευτή Λοροφίλη που από πλευρά της Χιλής ε, είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Χιλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές κύριε Πρόεδρε ότι για μας η Χιλή είναι μια χώρα παράδειγμα με την μεταπολίτευση και αυτή την εποχή προεδρεύει και στη Χελάκη που αντικατέστησε την προηγούμενη ομάδα. Εμείς πριν από λίγες μόνο μέρες, στο Κάντιθ, γιορτάσαμε τον κοινοβουλευτικό μας διάλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί την, ε, την επόμενη χρονιά στο Σαντιάγο της Χιλής. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, Πρόεδρε, διαπιστώνουμε τι δουλειά γίνεται για να προχωρήσουν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Είχα την ε, ευκαιρία να διαπιστώσω ότι το βασικό στοιχείο για να προχωρήσουν οι σχέσεις αυτές θα είναι η κινητοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Για πολιτικούς λόγους ενισχύθηκε ο διάλογος αυτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Χιλή ήδη από το 1984. για πολιτικούς λόγους επίσης θεσμοθετήθηκε η ομάδα του Ρίου το 1990 στην Ρώμη και για πολιτικούς λόγους επίσης ο πολιτικός αυτός ο υπουργικός ο διάλογος ε, προχώρησε το 1999 ακόμα πιο πολύ με το Ρίο Τζανέιρο. Τα γνωρίζετε όλα αυτά πολύ καλά εσείς λόγω της δικιάς σας προσωπικής πορείας. Σίγουρα ο πολιτικός αυτός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί και από δράσεις έτσι ώστε να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτής σύνδεσης που ολοκλήρωσε με την χώρα σας η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο. Επίσης, Πρόεδρε, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση στη Λατινική Αμερική. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί διάφορα. Έχει αποτύχει το σχέδιο ΑΛΚΑ, ορισμένες χώρες προτίμησαν διμερείς συμφωνίες, κατακαιρματισμός ε, της κοινότητας των Άνδεων, η Συμμαχία του Ειρηνικού, η Κίνα που ενισχύει τη θέση της ως εμπορικός εταίρος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μεταφέρεστε τις εντυπώσεις σας, πώς βλέπετε τις σχέσεις μας, πώς είναι και πώς θα έπρεπε να είναι με την προοπτική αυτή που έχουμε στα πλαίσια της νέας διάσκεψης κορυφής που θα έχουμε και την επόμενη συνεδρίαση της Eurolat πριν από την διάσκεψη της Eurolat. Ε, που θα γίνει λοιπόν στο Σαντιάγο της Χιλής. Ενημερώστε μας λοιπόν κύριε Πρόεδρε, πείτε μας τις απόψεις σας, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Σαλαφράγκα και καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ειλικρινά θαυμάζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι αυτό σημαίνει. Και όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο το κόσμο. Εδώ στο κοινοβούλιο αυτό ε, κανείς μιλάει, ε, υψώνει τη φωνή του, στηρίζοντας τη δημοκρατία, την ειρήνη, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα βήμα που έχει σαφείς απόψεις, που μιλάει με δυνατή φωνή, με σαφήνεια. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πάντα ήμουν φίλος των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Δεύτερον, Θέλω να σας πω δύο λόγια για την ε, Λατινική Αμερική. Είναι μια Ήπειρος όπου σήμερα ζουν 600 εκατομμύρια κάτοικοι. Είναι μια Ήπειρος που πέρασε τα πάντα. Ήταν ε, μια γενναιόδορη η χώρα, ε, χώρος μάλλον, με πάρα πολλούς φυσικούς πόρους, δεν είχε θρησκευτικά προβλήματα που είχαν σαν αποτέλεσμα να αλληλοσκοτώνονται λαοί στο όνομα του Θεού. Δεν είχε προβλήματα ρατσισμού που αντιμετώπισαν οι χώρες της Αφρικής. Παρόλα αυτά, με τόσο ευνοϊκές συνθήκες, τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας που ζούμε, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την υποανάπτυξη και την φτώχεια. Γι' αυτό λοιπόν η Λατινική Αμερική σήμερα έχει ένα χρέος απέναντι στον εαυτό της πρώτα απ' όλα και μια αποστολή να φέρει σε πέρας. Ο αιώνα αυτό θα πρέπει να είναι ο αιώνα τη αναγέννηση της Λατινικής Αμερικής. Και κατά κάποιο τρόπο το καταφέρνει η Λατινική Αμερική κατά το παρελθόν. Υπέφερε και ουσιαστικά ενίσχυε την ε, διεθνή οικονομική κρίση. Σήμερα όμως η Λατινική Αμερική είναι ήπειρος η οποία έχει αντιστηθεί περισσότερο, που έχει διατηρήσει την ικανότητά της για ανάπτυξη, για απασχόληση και παρόλο που έχασε την δημοκρατία, γενικευμένα θα έλεγα, σε ολόκληρο το χώρο αυτό τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 90, την ανάκτησε και πάλι και άρχισε να αντιμετωπίζει τις τεράστιες αυτές προκλήσεις που είχε μπροστά της. Χάρη στο δυναμικό που διαθέτει. Όμως ζούμε σε έναν αιώνα πολύ ιδιαίτερο. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια καταρρίφθηκαν τείχη και όχι μόνο του, της Ανατολής και της Δύσης που είχε το συμβολισμό μέσα από το τείχος του Βερολίνου. Υπήρχαν και άλλα τείχη όμως, βορρά νότου, του πλούτου και της φτώχειας δηλαδή. Ο βοράς ήταν ο πλούτος και ο Νότος η φτώχεια. Ε, δεν υπάρχει πια αυτό το τείχος. Υπάρχει όμως ε, ένα άλλο, το οποίο θα οδηγήσει στη πιο σημαντική ε, επανάσταση. Γιατί είναι μια επανάσταση της νέας κοινωνίας, που είναι η κοινωνία της πληροφορικής, με την γνώση και την πληροφορία να φτάνει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Είτε πρόκειται για την γεωργική επανάσταση λοιπόν, είτε για τη βιομηχανική. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά αντιμετωπίζουμε, και η χώρα μου ιδιαίτερα χιλή, μία πρόκληση που ήταν η πιο φτωχή απικία της Ισπανίας. Και σήμερα έχει μπροστά της μια τεράστια αποστολή και φιλόδοξη. Η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε τη χώρα μας. Πριν τελειώσει η δεκαετία αυτή, με μια αναπτυγμένη χώρα χωρίς στοχούς. Όταν θέσαμε το στόχο αυτό και την αποστολή αυτή, ξέραμε ότι τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουμε θα ήταν τεράστια. Και όντως, ήδη πριν από δύο χρόνια είχαμε τον ε, πέμπτο χειρότερο σεισμό που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. Ένα σεισμός με τεράστιες καταστροφές. Η Χιλή έχασε ένα στα τρία σχολεία ένα στα τρία νοσοκομεία που καταστράφηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όπως και ολόκληρη υποδομή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και παρόλο που ο κόσμος έμπαινε σε βαθιά κρίση, γιατί η οικονομική παγκόσμια κρίση ξεκίνησε το 2008 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα βέβαια, δεν έχει τελειώσει, εσείς οι Ευρωπαίοι το γνωρίζετε πολύ καλά, κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν παρόλα αυτά έθεσε ως στόχο και πρόκληση μπροστά της η Χιλή να πετύχει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, σε 10 χρόνια δηλαδή, να είναι η πρώτη, μακάρι και η μοναδική χώρα της ε, Λατινικής Αμερικής να καταφέρει να βγει από 200 χρόνια υποανάπτυξης, από 200 χρόνια συνύπαρξης με τη φτώχεια. Και για να τα καταφέρουμε αυτό βάζουμε επιμέρους σημαντικούς και φιλόδοξους στόχους. Πρώτα απ' όλα ανάπτυξη, δημιουργία απασχόλησης. Να αποτελέσουμε και εμείς μέρο του κόσμου, να ενισχυθούν οι επενδύσεις, οι εξαγωγές. Και ευτυχώς και παρά τις ε, δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε λόγω της οικονομικής κρίσης, της παγκόσμιας και του σεισμού, παρόλα αυτά προχωράμε και έχουμε πετύχει πολλά. Δημιουργούμε απασχόληση, αρκετή απασχόληση για να μπορέσουμε να απαλείψουμε την ανεργία, αλλά να μπορέσουμε και να ενισχύσουμε τομείς οι οποίοι δεν συμμετείχαν στον χώρο της εργασίας, οι πιο ευάλωτοι τομείς δηλαδή, οι γυναίκα συμμετέχουν στην ε, εργασία πολύ περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η οικονομική ισορροπία. Έτσι λοιπόν ε, βαδίζει ε, σε, με στέρεα βήματα η χιλή. Πρόκειται για μια ανάπτυξη η οποία είναι ισχυρή. Έχουμε οικονομικές προκλήσεις μπροστά μας. Έχουμε και κοινωνικές όμως προκλήσεις να μειώσουμε τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία της Χιλής. Τα πρώτα τέσσερα χρόνια που έχω εγώ την ηγεσία της κυβέρνησης, αυτό το θέσαμε σαν βάση για να αποτελέσει η Χιλή μια αναπτυγμένη χώρα, πριν τελειώσει η δεκαετία. Προχωρούμε λοιπόν και σε αυτό το τομέα. Όντως, ε, η φτώχεια μειώνεται, οι ανισότητες μειώνονται, έχουμε αναδιορθώσει σε βάθος ε, το κοινωνικό μας ε, πρόγραμμα και κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Χιλή, μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στην υγεία και στις κοινωνικές πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι η Χιλή είχε τους ε, βασικούς πυλώνες, δηλαδή σταθερή δημοκρατία, και πάντα στην ιστορία της σχεδόν έζησε η Χιλή με δημοκρατία. Υπήρξε μια διακοπή τη δεκαετία του 70 και του 80, ανέκτησε όμως τα τέλη της δεκαετίας του 80 τη δημοκρατία της Χιλή και είναι ο φυσικός τρόπος ζωής για τους χιλιανούς. Πέρα λοιπόν από μια σταθερή ε, οικονομία θέλουμε και μια ε, κοινωνική διάσταση μέσα σε ένα κράτος που να λειτουργεί καλά. Αυτή είναι οι βασικοί πυλώνες που είχαμε και την κοινωνική διάσταση και τη δημοκρατία. Θέλουμε όμως να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα και να συμμετέχουμε και εμείς ε, μεταξύ των χωρών του πρώτου κόσμου, με ειρήνη, με δημοκρατία, με ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε και νέους πυλώνες. Νέους πυλώνες που είναι τέσσερις βασικά και ολόκληρη η Λατινική Αμερική και οι Χιλή αυτούς τέσσερις πυλώνες είχαμε μείνει πίσω. Και ποιοι είναι αυτοί. Πρώτον, μεγάλη βελτίωση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, δίνοντας σημασία στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και γι' αυτό κάνουμε και τη μεταρρύθμιση της παιδείας. Ένα ποιοτικό άλμα επίσης όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία. Διότι ε, εμεί διπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό. Τεράστια προσπάθεια για να προωθήσουμε την καινοτομία και την γνώση, που είναι βασικά στοιχεία ε, χωρίς τέλος που ενισχύουν την ανάπτυξη. Επίσης, ε, περισσότερη ισότητα με λιγότερες αδικίες και λιγότερη φτώχεια. Αυτοί είναι νέοι πυλώνες, ε, λοιπόν, που θα μας επιτρέψουν, αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, να κάνουμε τη Χιλή μια χώρα η οποία να είναι ανεπτυγμένη και η οποία να απαλείψει την ένδια και να ζήσει σε ειρήνη και δημοκρατία. Και Εκεί βασίζονται και οι σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Χιλή ξεκίνησε τις σχέσεις της στη δεκαετία του 60 με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ευρωπαϊκή εμπειρία. Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, τόσο σκληρούς, θανατηφόρους, άγριους, η Ευρώπη κατάφερε να βγει από τη λογική της γραμμής Μαζινό και να πάει στην λογική της συνεργασίας και της ειρήνης. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Και γι' αυτό δόθηκε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Αυτή ήταν η λογική. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε τις σχέσεις της τότε με την τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, η Χιλή, και είχαμε μια συμφωνία συνεργασία για ελεύθερο εμπόριο, αλλά συνεργασία και σε άλλους τομείς, ε, την πολιτική, τον πολιτισμό. Πολύ καρποφόρα συνεργασία. Η Ευρώπη ήταν η ο πρώτος επενδυτής ε, στην Χιλή και ο πρώτος εμπορικός ε, εταίρος μετά την Κίνα. Και δίχως άλλο αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Η Χιλή όμως ήθελε και ένα άνοιγμα στον κόσμο και γι' αυτό ήθελε να δώσει σημασία και σε έναν άλλο πυλώνο που, πυλώνα που είναι να ενταχθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα περισσότερο από ό,τι το είχε πετύχει μέχρι τώρα. Έχει εμπορικές σχέσεις με 60 χώρες, με την Ευρώπη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κορέα. Σήμερα δουλεύουμε πάνω σε δύο νέες πρωτοβουλίες που είναι η Συμμαχία του Ειρηνικού όπου συμμετέχουν χώρες της Αμερικής όπως το Μεξικό και η Κολομβία αλλά και Χιλή που βλέπουν προς τον Ειρηνικό με πιο ενισχυμένη συνεργασία από την παραδοσιακή για εμπόριο αγαθών υπηρεσιών αλλά και επενδύσεις και ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Λίγο πολύ ακολουθούμε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι βέβαιο ότι η Λατινική Αμερική παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε είναι έναν αιώνα χωρίς πολέμους. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε την ολοκλήρωση που κατάφερε η Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν και θέλουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση μέσα στον κόσμο με ελεύθερο εμπόριο, με πολυμερείς, διμερείς, ε, συμφωνίες, δασμολογικές κλπ. Και έτσι να έχουμε μια χώρα πραγματικά ολοκληρωμένη σε ολόκληρο τον κόσμο με 75% ε, του ΑΕΠ να έρχεται από το εμπόριο πέρα όμως από τις οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις και τις κοινωνικές έχουμε δεσμευτεί και για πολιτική μεταρρύθμιση. Με αλλαγές στο θεσμικό τομέα, με ένα σύστημα σε θελοντική βάση ψηφοφορίες, από 8 εκατομμύρια έχουμε 13 εκατομμύρια τώρα πολίτες με δικαίωμα ψήφου και έχουμε υποσχεθεί και μεταρρύθμιση στα πολιτικά κόμματα όπως επίσης και για το εκλογικό σύστημα. Χώρα λοιπόν που αντιμετωπίζει τα διάφορα μέτωπα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά που θέλαν οι πατέρες μας αλλά που δεν κατάφεραν ε, ποτέ, δηλαδή αντιμετώπιση της υποανάπτυξης πρώτα απ' όλα. Θα ολοκληρώσω την ομιλία μου λέγοντα σα το εξή. Μάθαμε πολλά από την Ευρώπη, διδαχτήκαμε πολλά, γιατί στην Ευρώπη έχετε μια κοινότητα όχι μόνο ιστορική σημασία. Εμεί έχουμε δύο γλώσσε. τα πορτογαλικά και τα ισπανικά στη Λατινική Αμερική. Γιατί, γιατί ήμασταν απικία τη Ισπανία και τη Πορτογαλίας. Συνεπώ υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια η οποία διευκολύνει την ολοκλήρωση. Όμω αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης προς το παρόν στη Λατινική Αμερική δεν έχει γίνει τόσο σε βάθο όσο θα έπρεπε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεσμευτήκαμε με την ε, συμμαχία του Ειρηνικού, με σχέσεις με το Περού και άλλες, να προχωρήσουμε σε ολοκλήρωση και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη στον κόσμο. Επίσης δουλεύουμε και στο Trans-Pacific Partnership, που είναι ένα άλλο πρόγραμμα για μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών η πιο μεγάλη του κόσμου. Όπως κάποτε η Μεσόγειος ήταν ε, το κέντρο του κόσμου κάποτε, μετά ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός ίσως είναι η επόμενη ζώνη με τέτοιο δυναμισμό που να έχει την ίδια τύχη. Η Λατινική Αμερική και η Κεντρική Αμερική μπορούν να το πετύχουν αυτό. Γι' αυτό και είμαστε δεσμευμένοι υπέρ της ε, ολοκλήρωσης και με την Ευρώπη και γι' αυτό και θέλαμε τόσο πολύ την Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρώπη που έχει μια ρήτρα που λέει ότι θα ενισχυθεί η ολοκλήρωση αυτή τα επόμενα χρόνια, μετά από έξι χρόνια. Μέχρι τώρα μας έχετε υποδεχτεί πάντα τόσο καλά εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλο που δεν μπορώ να πω ακριβώς και το Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να τους καλέσουμε, θέλουμε μάλλον πρόσκληση σας 27 χώρες, εμείς είμαστε 33 χώρες, 600 εκατομμύρια κάτοικοι, ελπίζουμε τον Ιανουάριο που στη χώρα μας, στο Σαντιάγο της Χιλής θα γίνει η επόμενη διάσκεψη, αυτή θα πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να καταλάβουμε ότι μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης υπάρχουν και ιστορικοί δεσμοί, αλλά όχι μόνο ιστορικοί δεσμοί βάσει αξιών. Γιατί είμαστε μια κοινότητα οραμάτων και πρέπει να ενισχύσουμε την διαδικασία συνεργασίας μας και να αντιμετωπίσουμε μαζί την παγκόσμια πρόκληση μέσω μιας αναδιάρθρωσης του νομισματικού ή δημοσιονομικού συστήματος. Όλοι γνωρίζουμε, η Παγκόσμια παγκοσμια τραπεζα Ηνωμένες Πολιτείες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν τέτοιες αλλαγές. Άρα υπάρχει σύμπτωση απόψεων όπως διαπιστώνουμε από τις συνομιλίες που έχουμε και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, μάλλον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρώπης δηλαδή, αλλά και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τις δυνάμεις μας από κοινού για να πετύχουμε τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο κόσμος για να μετοπιστούν οι προκλήσεις, οι νέες δυσκολίε που έχουμε μπροστά μα να αντιμετωπίσουμε. Τελειώνει υπενθυμίζοντα σας κάτι που είπε ένας μεγάλο πολιτικός Αμερικανός που είπε ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι στον κόσμο. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν πώς έχουν τα πράγματα και βασίζονται σε αυτό και αυτοί που ονειρεύονται για το πώς θα θέλανε να έχουν τα πράγματα και προ τα εκεί οδεύουν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής για να αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την εικόνα που μας έχετε δώσει για τη χώρα σας, το πανόραμα της Λατινικής Αμερικής και των σχέσεών μας. Επίσης θα προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές. Έχω εννέα εγγεγραμμένους στον κατάλογο, βέβαια είναι περιορισμένος ο χρόνος μας γιατί η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει μια φορτωμένη ημέρησια διάταξη. Θα σας παρακαλέσω να είστε συντομότατοι, να παραμείνετε σε 1,5 λεπτό μέγιστο χρόνο αγόρευσης. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Κορέα Κάμπο, που είναι ο πρόεδρο μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Χιλή. Ευχαριστώ. Εξοχότατε κύριε Σεμπαστιάν Πινιέρα. Είναι για μας μια μεγάλη τιμή να σας δεχτούμε σε αυτό το σπίτι της δημοκρατίας στην Ευρώπη σε ένα χρόνο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής και φυσικά είναι και το έτος του, είναι η δέκατη επέτειος από τον Νοέμβριο του 2002 της πρώτης συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής. Θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο ε, Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μορένο, τον κύριο Λορενζίνο, τον κύριο Σαλαφράγκα φυσικά από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κύριο Άπλγκριν. Επίση, θέλω να χαιρετήσω όλου του καλεσμένου από την χιλιανή πλευρά και τελικά όλου του συναδέλφου, <clears throat> του Ευρωπαίου κοινοβουλευτικού που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή. Ω πρόεδρο τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τη Χιλή παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή τι εξελίξει που προκύπτουν για αυτή τη συμφωνία σύνδεσης είχα την τιμή μαζί με τον ομολογό μου τον Παύλο Λορεντσίνη να προεδρεύσουμε τη Μικτής κοινοβουλευτική Επιτροπής όπου γίνεται και η αξιολόγηση της προόδου στον τομέα της σύνδεση των δύο πλευρών. Η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να μην έχει νομοθετικέ αρμοδιότητες αλλά είναι μια φωνή που τα υπόλοιπα όργανα της Συμφωνίας Σύνδεσης ακούνε με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και αυτό δείχνει την ευθύνη που έχουμε αναλάβει ως κοινοβουλευτική. Οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί στους κύριους τομείς που διέπει η Συμφωνία αυτή της Σύνδεσης είναι προφανής και αρκεί να κοιτάξει κανείς την ταχεία αύξηση του εξωτερικού εμπορίου μεταξύ Χιλής και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δίνει μια ιδιαίτερη ευθύνη σε κάθε μία από τις πλευρές και καταδεικνύει και την ε, οριμότητα και τη θέληση πρόοδου για μια εδραίωση των στόχων που υπάρχουν στη Συμφωνία Σύνδεσης. Προφανώς θα υπάρχουν τομείς όπου η πρόοδος να είναι πιο περιορισμένη. Υπάρχει και η ανάγκη περαιτέρω εξέλιξη σε ορισμένους τομείς. Αλλά η πρόοδος ιδίως στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας ήταν ιδιαίτερα θετική και ελπιδοφόρα. Φαίνεται να υπάρχουν προοπτικές επίσης σε σχέση με την συνεργασία για τα ενεργειακά θέματα, ιδίω τα δίκτυα διανομής ενέργειας και τις ανανεώσιμες ενέργειες, όπου μπορεί να υπάρχει αμοιβαίο όφελος. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την παρουσία του Προέδρου Πινιέρα, ο οποίος έχει προεδρεύσει με υποδειγματικό τρόπο την κοινότητα ΣΕΛΑΚ των χωρών της Αμερικής και των χωρών της Καραϊβικής και που έχει προωθήσει όλο το έργο το οποίο έχει λάβει η χώρα στην Ένωση αυτή και το οποίο θα κορυφωθεί τον Ιανουάριο του 2013 με την πρώτη διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΣΕΛΑΚ στο Σαντιάγο της Χιλής. Η Χιλή έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αυτή και αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματο των σχέσεων μεταξύ λατινοαμερικανικών χωρών και Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορέσει με τον τρόπο αυτό να θεσμοποιήσει μια στρατηγική μεταξύ των δύο αυτών περιφερειακών ε, οντοτήτων και τα κοινοβούλια της Λατινικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και δεν έχουν φυστεί προσπαθειών μέχρι στιγμής για να δρεώσουν και την κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να συνοδεύει αυτή τη σχέση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο πρόεδρο Κορέα Ντεκάμπος. Δίνω το λόγο στον στο επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ κύριε στον κύριο Μιλαντεμόν. Συγγνώμη. Κύριε Πινιέρα και εγώ θέλω να προσθέσω τις δικές μου ευχές σε αυτές του κυρίου Σαλαφράγκα και του κυρία Κορέα Ντεκάμπους. Είναι σημαντική η παρουσία σα για την ευρωπαϊκή πλευρά τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων. Θα ήθελα να σα ζητήσω πώ εκτιμάτε τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα μάλλον της εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής. Βέβαια, αντλώ το συμπέρασμα από τα λεχθέντα σας ότι ήδη θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ θετική αυτή η συνεργασία, κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα στην Επιτροπή Εξωτερικών θεμάτων και φυσικά και ως Ισπανός επιθυμώ διακαώς να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και να εντατικοποιηθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Χιλή το των μάλλον, όσον ο Ειρηνικός φαίνεται να είναι πια η νέα περιοχή αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα πάρει την σκητάλη από τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Αυτό μας οδηγεί στο να θέλουμε να αντικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τη Λατινική Αμερική. Αναφερθήκατε σαν <clears throat> ένα σημαντικό στοιχείο την καινοτομία για την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα σας. Στον οικονομιστή διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σε σχέση με το πρόγραμμα που θέλετε να ξεκινήσετε, τα λεγόμενα startups, τις νέες εταιρείες οι οποίες δημιουργούνται, όπου θέλετε να προσελκύσετε και νέους επιχειρηματίες. Αυτό είναι κάτι πολύ καινοτόμο, αν δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, που υπάρχει πρόβλημα με το επιχειρήν και πρόβλημα με την απασχόληση. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λιγάκι καλύτερα τι περιέχει αυτό το πρόγραμμα, το startup, το οποίο είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα και το οποίο μπορεί να βελτιώσει το επιχειρήν στη χώρα σας. Η κυρία Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, μια μεγάλη ευχαρίστηση και για μένα να σας υποδεχτώ εδώ και να ακούσω τα λόγια σας και παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις προκλήσεις που θέτει στον εαυτό της η Χιλή, το θέμα της ισότητας όλων των πολιτών, την εξάλληψη της ένδυας. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για τις προσπάθειες που κάνετε για την ενσωμάτωση των πιο ευάλωτων πληθυσμών, ιδίως των Ιθαγενών πληθυσμών Μαπούτσε, Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μέσα στην κοινότητα αυτή του ειρηνικού πώς βλέπει η Χιλή τις ε, εντάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας για το σύμπλεγμα το νησιωτικό αυτό το οποίο διαμφισβητείται αυτή τη στιγμή από τις δύο χώρες. Με ποιο τρόπο λοιπόν η Χιλή θεωρεί ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο μέσα στην εταιρική σχέση του ειρηνικού. Επίσης έχετε κρατήσει ένα πάρα πολύ ενεργό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη, ένα πολύ θετικό ρόλο. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να αναδιαρθωθούν οι περιφερειακοί οργανισμοί χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα και οικονομικού χαρακτήρα όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά ποια είναι η άποψη της Χιλής σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όταν βλέπουμε τα διέξοδα στα οποία βρίσκεται το Συμβούλιο Ασφαλείας σε καταστάσεις όπως αυτή της Συρίας που υποσκάπτουν και την αξιοπιστία του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την θαυμάσια ε, ομιλία σας. Είμαι ο καθηγητής ε, Παναγιώτοφ από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Έχω εργαστεί στο παρελθόν στη Χιλή Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να μην ακούγεται καν η λέξη κρίσης στην ε, Χιλή. Τι μέτρα έχετε λάβει εσείς και η κυβέρνησή σας ώστε να είναι τόσο θετική η οικονομική κατάσταση στη Χιλή όπως είναι σήμερα. Eh, Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτοφ, κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά της Πράσινης Ομάδος και ε, Ελεύθερης Συμμαχίας. Έχετε παρουσιάσει με πολύ θετικό τρόπο τις πρόοδους που έχει επιτύχει η Χιλή και είσαστε πράγματι ένα άτομο το οποίο ονειρεύεται να επιτύχει περισσότερο. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι να εδρεωθεί στη Χιλή μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Σε σχέση με την Ευρώπη, όπου έχει επιτευχθεί αυτό με μια εστίαση όχι μονάχα σε την, στην εξορρυκτική οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγή βασικών προϊόντων, ένα από τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι η προστέμενη αξία που έχει δώσει στα προϊόντα αυτά. Η Χιλή ακόμα εξάγει βασικά προϊόντα όπως είναι προκυπευτικά, ε, αμπελουργικά προϊόντα τα οποία είναι ήδη κατά κάποιο τρόπο μεταποιημένα όπως είναι ο ίνος, ε, ορυκτά προϊόντα επίση, με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι μπορείτε να προχωρήσετε περισσότερο ώστε να έχετε μια μεταποιητική δραστηριότητα που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεταξύ του πληθυσμού. Και μίλησατε σε σχέση με την διάσκεψη κορυφή που θα λάβει η χώρα στην ε, Χιλή, όπου η αιστεία ήταν περισσότερο στα θέματα των επενδύσεων. Τι είδου επενδύσει θέλετε να προκρίνετε, Γιατί υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα επενδύσεων που μπορεί να υπάρχουν επενδύσεις παραγωγικές, επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα, επενδύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τέλος στις τελευταίες ε, διασκέψεις ε, κορυφής υπήρξε η συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών στην ε, Ήπειρο της Αντικής Αμερικής, στην Γουατεμάλα, στο Μεξικό και αλλού. Εσείς συμμερίζεστε την άποψη που έχει συζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το θέμα αυτό της βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να εγγραφεί και στην τελική διακήρυξη αυτής της διάσκεψης. Ευχαριστώ κύριε Λούνατσεκ. Ο κύριος Κόσουσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χάρηκα για την ε, παρέμβασή σας ιδιαίτερα. Μιλήσατε για τα τείχη τα οποία κατέρευσαν που χώριζαν τον κόσμο από ανατολικά δυτικά ή από βόρεια σε ερώτια ε, και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ προέρχομαι από την Τσεχία, από την Πράγα. Ζήσαμε κι εμείς την ε, κατάρρευση του, των τείχων. Προέρχομαι από ένα συντηρητικό κόμμα. Ορισμένοι λένε ότι είμαστε αντιευρωπαίοι, αλλά εδώ θα ήθελα να διορθώσω αυτή την λανθασμένη εικόνα για την πολιτική μας ομάδα. Έχουμε πολύ καλές εμπειρίες ως χώρα της Κεντρικής Ευρώπης με την ε, ολοκλήρωση της Ευρώπης και με την επίτευξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Γι' αυτό παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλη τη διαδικασία ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική και έχετε την απόλυτη υποστήριξή μα. Ευχαριστώ κύριε Κοσούσικ. Κύριο Πρέιό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή κάποια ερωτήματα τα έχουν θέσει οι συναδελφοί μου, θα σταθώ μονάχα σε ένα-δύο. Το κοινοβούλιο μας όπως είπατε, θέλει να είναι ο υπέρμαχος των ελευθεριών και της δημοκρατίας. Το 1997 ε, υποστήριξε την έννοια των, ε, της ιδιοκτησίας ορισμένων περιουσιακών στοιχείων στη Χίλη και αυτό, ε, αυτά τα θέματα είναι ακόμα επίδικα στην, ε, στη Χίλη. Ε, θα μπορέσετε εσείς να με διαβεβαίωσετε ότι μετά από τη δικαστική απόφαση θα επιστρέψουν αυτά τα άγαθα στον νόμιμο κατοχό τους, κυρία να έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πινιέρα. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς ο ίδιος σε σχέση με την θετική οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η Χίλη και το ερώτημα μου είναι το εξής. Τη στιγμή που υπάρχει η διεκδίκηση του λαού στους δρόμους για περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την γνώση, την εκπαίδευση των χιλιανών, θα προχωρήσετε σε νέες μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτικό τομέα και φυσικά και στον υγειονομικό τομέα. Γιατί φαίνεται ότι όλο και περισσότερο μειώνονται οι αποστάσεις γεωγραφικές, αλλά ε, αυξάνεται το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ένα άλλο συγκεκριμένο θέμα Αναφερθήκατε στο θέμα των οραμάτων, των οραμάτων για το μέλλον. Ε, για τη δικαιοσύνη όμως υπάρχει και εκεί ένα όραμα. όραμα. Υπάρχει περίπτωση του Καρμέλο Σόρια. Πέρσι η, η Ισπανία ζήτησε να συλληφθούν έξι αξιωματικοί του χιλιανού στρατού για αυτό το αδίκημα. Θα συνεργαστεί η χιλιανή δικαιοσύνη για να μπορέσει να υπάρξει δικαιοσύνη στην περίπτωση του Καρμέλο Σόρια ή όχι. Κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κοινωνία των πολιτών της χώρας σας, η οποία εκπροσωπείται και από τους Μαπούτσε και από τους φοιτητέ που ήρθαν, είναι μια κοινωνία των πολιτών η οποία μας μεταφέρει κάποιες ιδέες κάπως διαφορετικές από αυτές που μας αναφέρατε εσείς. Ιδέες που μιλούν για τον κοινωνικό αποκλεισμό και για τις διακρίσεις. Ε, βέβαια η χώρα σας πέτυχε τα τελευταία χρόνια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Οι εμπορικές σας σχέσεις ε, διευρύθηκαν σε διεθνές ε, επίπεδο, αλλά συγχρόνως υπάρχει ένα χάσμα, γιατί υπάρχει μεγάλη φτώχεια ιδιαίτερα στις κοινωνίες των Μαπούτσο στον Νότο. Επίσης γίνονται πολλές παραβιάσεις που μένουν ε, χωρίς κυρώσεις, χωρίς τιμωρία. Έγινε απεργία πείνας πρόσφατα από τους Μαπούτσο ακριβώ για αυτό το θέμα και σας έχω στείλει και σχετικά επιστολή. Γίνεται επίσης μεγάλη συζήτηση για τον νόμο για την αλία μικρής κλίμακας. Υπάρχει κινητοποίηση των ε, αλλιέων γιατί δεν ζητήσατε την γνώμη τους για το νόμο αυτό. Υπάρχει νομοθεσία Πέσκερ που έχει το όνομα του Υπουργού σας που περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και τις ελευθερίες των ατόμων. Τέλος, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό υπάρχουν πολλοί βουλευτές που ανησυχούν ιδιαίτερα για την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά του Μαπούτσου κάτι το οποίο έφτασε και στη UNICEF. Είναι τροπή να υπάρχει τέτοια παραβίαση. Εμείς ε, ενημερώσαμε σχετικά και την κυρία Στον. Το να δοθεί σημασία στην ε, βελτίωση, στην ενίσχυση της δημοκρατίας και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας, την οποία χώρα σας εμείς αγαπάμε και εννοείται ότι σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας για αυτή την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού των Μαπούτσε και ιδιαίτερα σας ε, να ξέρετε ότι εμείς εδώ δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτά και θα παρακολουθούμε το τι κάνετε. Θέλουμε να τους ε, ακούσετε κι εσείς όπως τους ακούμε εμείς εδώ. Ευχαριστούμε κυρία Μιράντα και κυρία Μούνιεθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πινιέρα, κύριε Πρόεδρε Πινιέρα, είναι τιμή για μας που σας έχουμε εδώ και να μας ε, παρουσιάσετε τα θέματά σας, όπως είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και στα πλαίσια της δικιάς μας ε, Επιτροπής για τις Σχέσεις μας με τη Χιλή στην ε, χώρα σας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπα. Την αλήθεια ότι μας ενώνουν οι τεράστιες επενδύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Χιλή, η σημασία που δίνουμε Πέρα από τα συγχαρητήρια που θέλω να σας δώσω, θέλω να υπενθυμίσω ότι ήταν ιστορική σημασία η εκλογή σας όσον αφορά την μεταπολίτευση στη Χιλή. Θα σας υπενθυμίσω κάτι και θα σας ρωτήσω και μερικά πράγματα. Η Παγκόσμια Τράπεζα αυτή τη εβδομάδα παρουσίασε έκθεση όπου φαίνεται ότι το 12% του πληθυσμού της Χιλής, 2 εκατομμύρια περίπου δηλαδή, έχουν μπει τώρα στη μεσαία τάξη στη Χιλή. Το αντίθετο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου υπάρχει η αντίθετη διαδικασία, δηλαδή ότι η μεσαία τάξη κατεβαίνει. Το αντίθετο λοιπόν συμβαίνει στην ε, Χιλή. Παραμένουν όμως ανισότητες, όπως υπενθύμησαν κάποιοι συνάδελφοι. Και οι πολίτες και στην Ευρώπη αλλά και στην Χιλή ζητούν μεταρρυθμίσεις. Στη Χιλή για την εκπαίδευση για παράδειγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από το κράτος για να ενισχυθεί η ευημερία στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποίησης και της υγείας και της εκπαίδευσης. Τώρα, οι επόμενες εκλογές θα είναι οι πρώτες όπου θα συμμετέχουν και οι χιλιανοί που δεν ζουν στην Χιλή και που δεν είχαν αυτό το δικαίωμα μέχρι τώρα. Αυτό θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Στα πλαίσια της εξωτερικής τώρα πολιτικής της Χιλής ξεχωριστικό ρόλο για να λυθούν περιφερειακές συγκρούσεις. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση με την Παραγουάη που έχει μείνει απομονωμένη. στον ε, χώρο. Κάνει κάποιες προσπάθειες η Χίλη προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μονίθ. Τελευταίος ο κύριος ε, Πάφες. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κύριος Καρσές Ραμών. Πώς βλέπει η κυβέρνηση της Χιλής σήμερα τις συγκρούσεις στην ε, θάλασσα ή και όχι στη θάλασσα με τη Βολιβία. Υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις ιστορικά. Και εμένα, ε, εγώ μάλλον προσέχω ιδιαίτερα την περίοδο 70-80, αναφερθήκατε και εσείς κύριε Πινιέρη και είπατε ότι διακόπη δημοκρατία τότε. Στην Ευρώπη την περίοδο αυτή εμείς τη λέμε στρατιωτική δικτατορία, βία περίοδο σκληρή. Και εσείς λέτε απλώς ότι πρόκειται για μια περίοδο διακοπής της δημοκρατίας. Έτσι τη χαρακτηρίσατε αυτή την περίοδο στην ομιλία σας. Ευχαριστούμε. Λέει ο Πρόεδρος. Βλέπετε κύριε Πρόεδρε Πινιέρα πόσο πολύ ενδιαφέρονται οι ευρωβουλευτές μας ε, για τη χώρα σας. Το δείχνει και η παρουσία τόσο πολύ άριθμη των ευρωβουλευτών εδώ στην αίθουσα. Λοιπόν, απαντήστε μας. Σας ευχαριστώ, όντως μου κάνατε πολλές ερωτήσεις. Κάποιες είναι περισσότερο διαπιστώσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Το πρόγραμμα Startup Chile. Είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε για να ενισχύσουμε την ε, τεχνολογία και τις επιστήμες, διπλασιάζοντας τις επενδύσεις μας και ενισχύοντας την ε, γνώση. Θέλουμε να προσελκύσουμε ε, φορείς από όλο τον κόσμο στη Χιλή. Τους δίνουμε βίζα, τους επιτρέπουμε να εγκατασταθούν και τους επιδοτούμε κιόλας με 50.000 δολάρια για να μπορέσουν να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους στη Χιλή. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό έχει θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των επιστημών και της γνώσης στη χώρα μας. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει στεφθεί από επιτυχία. Είχαμε πάρα πολλές υποψηφιότητες από ολόκληρο το κόσμο. Ο καθένας τους πρέπει να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα καινοτομία και ε, τεχνολογίας. Η κυρία Γκόμες ε, με ρώτησε για τα κοινωνικά προγράμματα στην Χιλή και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους Μαπούτσε και στην Trans-Pacific ε, Partnership και τη θέση μας στα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, το κοινωνικό πρόγραμμα στη Χιλή. 70% των δημοσίων δαπανών πηγαίνουν σε κοινωνικές δαπάνες στη Χιλή για να μειωθούν οι ανισότητες, οι οποίες είναι πάρα πολλές ε, στη χώρα μου και για να μειωθεί η ένδια, που από 40% που ήταν το 90 έχει πέσει στο 14% σήμερα, που είναι το χαμηλότερο σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Βέβαια σημαίνει αυτό 2,5 εκατομμύρια χιλιανοί ακόμα που ζουν στη φτώχεια, που είναι πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε 16.000 ε, δολάρια κατά κεφαλή εισόδημα στη Χιλή, είναι ντροπή. Προσπαθούμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα επίση που στοχεύει ιδιαίτερα τι πιο φτωχέ οικογένειε. με τρει επιλόνες. Αξιοπρέπεια πρώτα απ' όλα. Αξιοπρέπεια που είναι ήδη πολύ βασικό. Ο δεύτερο πυλώνα είναι η υπευθυνότητα. Αν η οικογένεια αναλάβει κάποιε ευθύνε το να στέλνει τα παιδιά τη στο σχολείο για παράδειγμα, κάτι το οποίο ελέγχουμε, τότε παίρνει κάποια επιπλέον χρήματα. Και έπειτα υπάρχουν τα επιτεύγματα. Αν καταφέρει να βελτιώσει, για παράδειγμα, η οικογένεια το ε, επίπεδο εκπαίδευσης των ε, παιδιών τους, παίρνουν επίσης κάποια χρήματα. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για αρρωγή, έχει και στόχους. Βοηθάμε τις πιο φτωχές οικογένειες, εκείνες όμως που βάζουν και δικιά τους προσπάθεια για να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Τώρα για τους Μαπούτσε. Οι Μαπούτσι ε, βρίσκονταν στη Χιλή πολύ πριν από τους Ισπανούς. Δεν είναι οι Ισπανοί που ανακάλυψαν ε, την Αμερική, πολύ πριν είχε ανακαλυφθεί αυτή. Συνεπώς, μαζί τους, θα λέγω ότι έχουμε κάποιο χρέος. Νιώθουμε πολύ περήφανοι για την ιστορία τους. Και γι' αυτό και προωθούμε μια νέα πολιτική για αυτούς. Μια νέα μεταχείριση. Πρώτα απ' όλα, συνταγματικά αναγνωρίζουμε τον λαό αυτό. συμμορφωθήκαμε προ το ψήφισμα 169 του ΙΕ που λέει ότι πρέπει προηγουμένω να έχουμε ζητήσει τη γνώμη του για κάθε απόφαση που του αφορά κτλ. Έπειτα στην Αροκανία, στην περιοχή δηλαδή που ζει ένα μεγάλο μέρο του λαού αυτού, έχει δύο σχέδια από εμά. Ένα που είναι για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ένα άλλο που είναι για την αναβάθμιση και την ε, βοήθεια που δίνουμε για τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους κτλ. Πράγματα που αποτελούν και την ψυχή της χώρας μας. Τώρα, για την εταιρική σχέση του ειρηνικού. Έχουμε μια πρωτοβουλία για τις χώρες αυτές του ειρηνικού. Η Νέα Ισλανδία, η Σιγκαπούρη, το Μπρουνέι και η Χιλή συμμετέχουν. Και μετά ήρθαν και οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδά, το Περού και χώρες άλλε του ειρηνικού όπω το Βιετνάμ, η Αυστραλία, η Μαλαισία. Και έτσι δημιουργήθηκε μια ε, περιοχή ελεύθερων συναλλαγών η μεγαλύτερη του κόσμου. Έτσι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την αποτυχία του γύρου της Ντόχα. Όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείες, ναι, θέλουν αλλαγές. Και για τους ε, δημοσιονομικούς οργανισμούς, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ε, το θέλει, αλλά και η χώρα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι πρέπει όντως να υπάρξει μια διαφορετική πραγματικότητα Πρέπει να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα. Τώρα, για τον κύριο Παναγιώτοφ και τη Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Γιατί δεν μιλάμε για κρίση στη Χιλή. Κοιτάξτε, η κάθε χώρα ζει τη δικιά της κρίση που είναι διαφορετική από εκείνη της, ε, του γείτονα. Εμείς έχουμε κρίση επειδή, όχι λόγω ανεργίας, επειδή θέλουμε να μειώσουμε τη φτώχεια από την οποία υποφέρει η χώρα μας τα τελευταία 200 χρόνια. Έχουμε ανάπτυξη 6%, έχουμε αύξηση της απασχόλησης, οι επενδύσεις αυξάνονται δύο και τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι το ΕΠ μας. Συνεπώς, στην Κίνα δεν μιλάμε για την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά πώς θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την απασχόληση. Εμείς στην Χιλή μιλάμε για την κατανομή των κερδών, μιλάμε για την επιτάχυνση των προγραμμάτων μας και πώς θα ενισχύσουμε τα ωφέλη για τον πληθυσμό. Είμαστε σε μια κατάσταση διαφορετική βέβαια από αυτή της Ευρώπης, γιατί εμείς προχωράμε και θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα για τις επενδύσεις. Όντως είναι κάτι που έχουν κάνει πολλές κυβερνήσεις στην Χιλή και η δικιά μας βέβαια ακολουθήσαμε μια υπεύθυνη οικονομικά πολιτική με διαρθρωτική ισορροπία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν έχουμε ήλιο εξοικονομούμε για να αντιμετωπίσουμε τις σκοτεινές μέρες. Αυτό είναι ο νόμος. Είναι υποχρεωτικό για μας αυτό. Άρα αποταμιεύουμε όταν μπορούμε να αποταμιεύσουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρου αυτούς σε πιο δύσκολες μέρες. Και έτσι καταφέραμε να ε, ξεπεράσουμε την κρίση του 2009 και καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία παρά τη βαθιά αυτή κρίση που είναι η δεύτερη χειρότερη στον κόσμο οικονομικά μετά το 29 δεν πέσαμε σε ύφεση όπως είχε συμβεί στις προηγούμενες κρίσεις. Αλλά προχωράμε και επιπλέον γιατί κανείς στη ζωή παίρνει διδάγματα. Ότι δεν μπορούμε να ζούμε πάνω από τις οικονομικές μας δυνατότητες. Και η Χιλή ξέρει ότι κάποια στιγμή θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό και προετοιμάζεται γι' αυτό. Κάτι το οποίο δεν έγινε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ειδού οι συνέπειες. Να απαντήσω τώρα στην κυρία Λούνατσεκ. Για την εξαγωγή πρώτων υλών. Πράγματι, η Χιλή ε, βασίζεται πάρα πολύ στις πρώτες ύλες. Σε πολλά υλικά που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία. Ξέρετε ότι για παράδειγμα ο ίνος μας βελτιώνεται η ποιότητά του. Έχουμε και μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά και καλύτερη, ε, και καλύτερη ποιότητα και ποσότητα μεγαλύτερη. Η ξυλία επίσης βελτιώνεται. Και αυτό είναι πολύ βασικό και γι' αυτό και θέλουμε να προσελκύσουμε τεχνολογία και καινοτομία. Έχουμε τη Max Planck και άλλες εταιρείες που έχουν έρθει και μας προσφέρουν γνώση, επιστήμη, τεχνολογία, καινοτομία, γνώση. Όλα αυτά αυξάνουν την αξία των πρώτων μας υλών και άρα μας βοηθούν για φόρο ανάπτυξη. Και αυτό θα αποτελέσει και το θέμα της διάσκεψης που θα έχουμε της ε, ΣΕΛΑΚ την επόμενη χρονιά Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής. Θα μιλήσουμε για επενδύσεις αλλά για υπεύθυνε επενδύσεις, υπεύθυνε κοινωνικά επενδύσεις, υπεύθυνε περιβαλλοντικά επενδύσεις για να υπάρξει μια αϊφόρος, μια βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα της διάσκεψης κορυφής. Πώς δηλαδή θα αλλάξει η λογική της ανάπτυξης για να είναι πιο αρμονική από κάθε άποψη κοινωνική αρμονία, περιβαλλοντική αρμονία και οικολογική και η υπευθυνότητα όσον αφορά μια ανάπτυξη για όλους, που να επιτρέπει σε όλους τους κατοίκους όλων ε, των λαών και της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη αυτή και στο φέλη της. Τώρα στη Χιλή, όπω και σε πολλέ άλλε χώρε Λατινικής Αμερική, είναι αλήθεια ότι έχουμε πολύ ενδοοικογενειακή βία σε βάρο των γυναικών και των παιδιών πολλέ φορέ. Και γι' αυτό έχουμε κάνει τεράστιε αλλαγέ στην νομοθεσία μα. Ένα από του στόχου τη κυβέρνησή μα ήταν να παλευθούν όλε οι διακρίσει που μπορεί να υπάρχουν στον νόμο. Και όντω τα καταφέραμε για πολλέ. Νομικά δηλαδή τι απαλήψαμε. Γιατί οι πολιτιστικέ διακρίσεις δεν αλλάζουν με τον νόμο βέβαια, αλλάζουν με την οτροπία με τη στάση, με την παιδεία. Έτσι λοιπόν θέλουμε με την κυβέρνησή μας να φροντίσουμε να μην υπάρχει απολύτως κανένας νόμος που να ε, προσφέρει περιθώρια για διακρίσεις σε βάρος των γυναικών ή των παιδιών. Αλλάζουμε δύο νόμους επίσης τώρα που έχουν να κάνουν ε, με τις υγικές σχέσεις και ένας άλλος που λέει ποιος αναλαμβάνει το κόστος όταν δουλεύει και η γυναίκα. Έχουμε ένα Υπουργείο πάντω στη Χιλή που επικεντρώνεται σε αυτόν ακριβώ το στόχο. Έχουμε αυξήσει επίση τι κυρώσει. Όποιο ε, προχωράει σε βία σε βάρο των γυναικών, ιδιαίτερα όταν έχει συναισθηματική σχέση μαζί τη, τότε τιμωρείται παραδειγματικά. Και όντω έχουν μειωθεί οι περιπτώσει βία, ενδοικογενειακή ε, βία. Είχαμε πάρα πολλές και πιστεύουμε ότι ο αριθμός των περιπτώσεων αυτών θα συνεχίσει να μειώνεται. Έρχομαι τώρα στο θέμα της περίπτωση Κλαρίν. Πράγματι υπήρξε στην εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας απαλωτρίαση της εφημερίδας αυτής του Κλαρίν και οι κάτοχοί του ζήτησαν να υπάρξει αποζημίωση. Το θέμα αυτό ετέθηκε από ένα ε, Ισπανό πολίτη υπήκο, ο οποίο έθεσε το θέμα στα διεθνή δικαστήρια, η Χιλή σέβεται πάντα τι αποφάσει των διεθνών δικαστηρίων. Αν λοιπόν αποφασίσει ότι ούτω έχει το διεθνέ δικαστήριο, η Χιλή θα α, τηρήσει την απόφαση του δικαστηρίου και θα την εφαρμόσει, αλλά αυτό το οποίο ζητά το διεθνέ δικαστήριο και όχι αυτό το οποίο ζητά ο Ενάγων, αλλά το Ίδρυμα που, στρέφεται, που περιστρέφεται από τον κύριο Γκασέ και άλλους στην Ισπανία. Η χώρα μας λοιπόν σέβεται το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο και σέβεται πάντα την έννοια του κράτους δικαίου. Εν τέλει, η αίτηση για μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και στην υγεία. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι για να υπάρξει μια εκβάθρον μεταρρύθμιση. Έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό της ε, παιδείας από σχεδόν 9 δισεκατομμύρια σε 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό είναι μια τεράστια αύξηση γιατί ξέρουμε ότι δεν πρέπει μοναχά να αλλάξουμε την ποιότητα της ε, ε, εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, αλλά επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε και την πρόσβαση στην παιδεία σε όλο μας τον πληθυσμό. Για πρώτη φορά έχουμε ε, δεσμευτεί να υπάρχει δυνατότητα δωρεάν προσχολικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Έχουμε αυξήσει λοιπόν σημαντικά την ε, συμβολή του κράτους στην προσχολική εκπαίδευση και επίσης έχουμε βελτιώσει τα προγράμματα για υποτροφίας και για δάνεια για την ανώτατη εκπαίδευση. Τώρα, όλοι οι χιλιανοί φοιτητέ που έχουν ε, υψηλά προσόντα έχουν το δικαίωμα να έχουν μια υποτροφία και οι υπόλοιποι έχουν το δικαίωμα να έχουν δανειοδότηση με 2-3% και πληρώνουν μόνο από τη στιγμή που αρχίζουν να εργάζονται και μετά από 15 χρόνια εκπνέει το υπόλοιπο χρέο. Ο στόχο μα είναι λοιπόν να υπάρχει ισοδίκαια πρόσβαση στην πρόσβαση στην ε, παιδεία. Υπάρχει τώρα διαφορά απόψεων μεταξύ του κυβέρνηση και ορισμένων φοιτητών, αλλά η κυβέρνηση έχει εκλεγεί από μια απόλυτη πλειοψηφία του λαού τη Χιλή. Κάποιοι στη Χιλή λένε ότι πρέπει να είναι τελείω δημόσια η παιδεία. Εμεί δεν πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι πρέπει όλη η κοινότητα μαζί, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, να μπορούν να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για το λαό της Χιλής. Και αυτό αφορά από την προσχολική μέχρι την πανεπιστημιακή παιδεία. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι οι γονεί οι οποίοι αποφασίζουν για τα παιδιά του και οι νέοι οι οποίοι πρέπει να αποφασίζουν πού θα σπουδάσουν. Αυτή είναι μια βασική ενοιολογική διαφορά. Άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν η ανώτατη εκπαίδευση για όλους τη χειρή. Εμείς δεν θέλουμε με τα λεφτά των φορολογουμένων να πληρώνεται η παιδεία πανεπιστημιακή των ε, πλουσίων. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τις υποτροφίες και το σύστημα των δανείων που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και θετικό για τους νέους, ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά δεν θέλουμε τη δωρεάν παιδεία σε πανεπιστημιακό επίπεδο για όλους, γιατί αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φτωχών για τους πλούσιους, όταν ακόμα υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια χιλιανών που βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της ένδυας. Για την περίπτωση Καρμέλο Σόρια, εμεί φυσικά καταδικάσουμε όλε τι παραβιάσει στα ανθρώπινα δικαιώματα που λαμβάνουν στη Χιλή. Κατά την άποψή μα, δεν υπάρχει κανένα λόγο, δεν υπάρχει καμία συγκυρία, καμία, ε, κανένα αποχρόν λόγος που μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επειδή υπήρξαν κατά τη διάρκεια τη δικτατορία η στρατιωτική κυβέρνηση. Υπήρξαν φυσικά παραβιάσεις σοβαρές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο η χιλιανή δικαιοσύνη αντιμετωπίζει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η χιλή έφερε στην δικαιοσύνη με υποδειγματικό τρόπο όλους αυτούς οι οποίοι έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα συνεργαστούμε για να γίνει γνωστή η πραγματικότητα και να έρθουν ενώπιον τη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει τη νομοθεσία μα και βάσει τη συνθήκη τη Ρώμη, την οποία έχει, υπογράψει η Χιλή. Αυτά που είπε η κυρία Μιράντα. Ναι, υπάρχει, υπάρχουν διακρίσει στη χώρα μα, υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Εμεί εγκρίναμε τον νόμο κατά των διακρίσεων. Η πρώτη φορά που στη Χιλή υπάρχει νομοθεσία που καταδικάζει ανοιχτά κάθε είδου διακρίσει που είναι αυθαίρετε, υποχρεώνει το κράτο να εργαστεί εναντίον των διακρίσεων και δίνει εργαλεία σε αυτού οι οποίοι είναι υπέρμαχοι τη ισότητα για να αντιμετωπίσουν κάθε τύπο διακρίσεω. Από πολλέ απόψει, ο λαό των Μαπούτσε είναι θύμα διακρίσεων. Καταρχήν σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο βρίσκονται κάτω από το μέσον όρο τη χώρα μα και γι' αυτό το πρόγραμμα Ραουκανία προσπαθεί να του βοηθήσει. Στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι και το ερώτημα που θέσατε είναι σαφέ. ότι εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιαδήποτε συνθήκε. Για το νόμο περί αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα. Ο πρώτος στόχος αυτού του νόμου είναι να πάψουν να χάνονται οι θαλάσσιοι πόροι της Χίλης. Στη Χίλη η υπεραλίευση έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλά αλλιευτικά είδη. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, να καταστραφούν αυτοί οι αλληλευτικοί πόροι. Θέλουμε να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα. Αυτό φυσικά προσκρούει σε κάποια συμφέροντα. Ορισμένοι θέλουν να συνεχίσουμε την αλόγιστη αλίευση. Θέλουμε επίση να προστατεύσουμε του μικρού βιοτεχνικού αλεί, που είναι το 90% των αλίων στη χώρα μα, με το να του δώσουν τη δυνατότητα να έχουν το πρώτο μήλι από τι ακτέ μόνο για αυτού. Αλλά υπάρχουν και αλείς οι οποίοι δεν είναι βιοτεχνική αλία και οι οποίοι είναι περισσότερο βιομηχανικοί και οι οποίοι θα θυγούν από αυτό το νόμο και προσπαθούν να υποστηρίξουν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Ο καθένα μπορεί να έχει ένα συμφέρον, αλλά δεν αρκεί να είναι συμφέρον, πρέπει το συμφέρον αυτό να είναι δίκαιο. Η χώρα μα και η κυβέρνησή μα πρέπει να σεβαστεί το γενικό συμφέρον. Ήταν ένα πολύπλοκο ε, νόμο, συζητήθηκε στην ε, Γερουσία, στην, ε, στο κοινοβούλιο μα, όπου δεν έχουμε πλειοψηφία και ενεκρίθη και θα περάσει μετά στη, στη Γερουσία. Αν τελικά εγκριθεί λοιπόν από τη, τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα της Χιλής, τότε αυτή είναι η έκφραση του λαού μας. Ορισμένοι χρησιμοποιώντας τη βία θέλουν να υπερασπιστούν συμφέροντα που στρέφονται κατά του γενικού συμφέροντος. <clears throat> Όταν μιλάτε για ένα νόμο καταστολής, φαντάζομαι ότι μιλάτε για ένα νόμο ο οποίος έχει να κάνει με τη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους. Εγώ πιστεύω στην ελεύθερη έκφραση. Είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα. Δεν είναι ένα δώρο που δίνει η κυβέρνηση στους πολίτες. Είναι δικαίωμα των πολιτών. Συγχρόνως όμως είναι απαραίτητο να σεβόμαστε και τα δικαιώματα των υπολείπων. Και όχι με το πρόσχημα της ελεύθερης έκφρασης να υπάρχουν καταστροφές ε, περιουσίας ιδιωτικής ή δημόσιας ή να τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές άλλων ανθρώπων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίο να είναι συμβατό με την ελευθερία τη έκφραση και χωρί να βλάπτει κανένα. Εμεί ποτέ δεν έχουμε εμποδίσει μία ε, διαδήλωση κυρίω φοιτητών γιατί όλα αυτά ενταγιάται το σύνταγμα τη ε, Χιλή. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τη ζωή και την περιουσία των άλλων. Επίση, για το, αυτό που λέτε για τη μέση τάξη, πράγματι η μείωση τη ένδυα του τμήματο των ενδέων πολιτών από 40 σε 14% ήταν πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα όλων των κυβερνήσεων που ακολούθησαν την ε, επαναφορά της δημοκρατίας και οι οποίες ανήκαν και σε πολιτικές δυνάμεις αντίθετες από τη δική μου. Αλλά ο στόχος ήταν η ανάπτυξη της χώρας, η μείωση της ένδυας που όπως σας είπα από το 1990 στο 40% έχει φτάσει στο 14% αυτό είναι μια σημαντική αύξηση της μέσης τάξης στην χιλία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια κοινωνία που πιο στηρίζεται σε πιο στερεούς και σταθερούς πυλώνες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όλοι οι πολίτε να ψηφίζουν. Έχουμε περάσει ένα νομοθέτημα για τα, θέματα αυτά, για τα θέματα αυτά και ελπίζουμε ότι ακόμα και οι χιλιανοί που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν ένα δεσμό με τη χώρα μας θα μπορούν να συμμετέχουν στι εκλογέ. <clears throat> Τέλος. Μου είπατε για την το Είναι ένας νέος θεσμός ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο για την κρίση της δημοκρατίας στην Παραγουάη και επίσης σε σχέση με αυτό το οποίο έγινε στο Εκουαδόρ. Στις περιπτώσεις αυτές κινητοποιηθήκαμε αμέσω για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Ο φορέας λοιπόν αυτός έχει πετύχει αποτελέσματα, επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, ο κ. Γκασές με ρώτησε για τη Βολιβία καταρχήν. Είμαστε γείτονε με τη Βολιβία, έχουμε μια συμφωνία οικονομικής συνεργασίας και όπως ξέρετε έχουμε μια διαφορά ερμηνείας για τα δικαιώματα της, των δύο χωρών. Υπάρχει μια συνθήκη, η συνθήκη του 1904, και η οποία έχει κυρωθεί από τα αντίστοιχα κοινοβούλια. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί πάντα σε διάλογο με τη Βολιβία μέσα στα πλαίσια του σεβασμού της συνθήκης του 1904 και που, που διέπει τις σχέσεις μας μεταξύ μας. Μετά από την στρατιωτική, ε, για τη στρατιωτική δημοκρατία, ναι, στρατιωτική δικτατορία. Ναι, ήταν διακοπή της δημοκρατίας, ήταν μια στρατιωτική δικτατορία και υπήρξαν πράγματι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά έχουν περάσει ήδη πάνω από 40 χρόνια. Αυτό που θέλουμε στη Χιλή είναι, αντί να συνεχίσουμε να έχουμε εσωτερικούς διχασμούς, είναι να ξαναενωθούμε μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις και τα μεγάλα οράματα που έχουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε εμείς εδώ τη συνεδρίασή μας, αλλά προηγουμένως, Πρόεδρε, να σας πω πως ε, θέλω να υπενθυμίσω πως η δημοκρατική ρήτρα που περιλαμβάνουν οι συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες και που χαρακτηρίζουν και τις ε, σχέσεις μας μαζί τους, ξεκίνησε στον ε, κήπο των ε, πορτοκαλέων στην ε, Χιλή. Θέλω λοιπόν στη, στο Μέγαρο Μονέδα στην Χιλή. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλοι θέλουμε να αποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο από τις ρήτρε αυτές. Εμείς είμαστε υπέρ του δυναμισμού της Λατινικής Αμερικής. Όπως είπε και ο συνάδελφος Κορεντεκάμπο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πιέσουμε τα άλλα θεσμικά όργανα, ώστε να μπορέσουμε να αποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο από τη συμφωνία αυτή. Εσείς, ατυχώς αναφερθήκατε στη γραμμή Μαζινό, Πρόεδρε. Σήμερα, αντί για αυτήν την γραμμή Μαζινό, έχουμε την Ευρώπη χωρίς σύνορα. Όλοι μαζί Θέλουμε να ενισχύσουμε και τη συνεργασία μας με την χιλιόλυση. βρισκόμαστε εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι η Λατινική Αμερική δεν είναι περιφερειακός παράγοντας αλλά κεντρική σημασία παράγοντας. Και είναι πολύ βασικό και στη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και στον Ατλαντικό και στον ε, Ειρηνικό. Όντως, στην κοινοβουλευτική διάσκεψη θα έρθουμε στο Σαντιάγο της Χιλής. Θα συναντηθούμε μαζί σας, ελπίζουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό τον ανοιχτό και ε, καρποφόρο διάλογο που είχαμε μεταξύ μας και να σας ε, επαναλάβω ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στη σχέση μας. Ευχαριστούμε. Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Χιλή στην Αλβανία. Take up the next agenda item. Θα πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, το υπαριθμό 4, έκθεση πρόοδου 2012 για την Αλβανία. Είναι η δεύτερη συζήτηση στον αφορά το σχέδιο εκθέσεων την Αλβανία Πρώτη συζήτηση έχει γίνει για προτάσει ψηφίσματος για τις χώρε διεύρυνση. Να επενθυμίσω στου συναδέλφου, όλη την έκθεση προόδου για το 2012 Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τις προόδους που έχει πετύχει η χώρα και πρότεινε να της δοθεί καθεστώς υποψήφιας χώρας με την επιφύλαξη της ολοκληρώσεως βασικών μεταρρυθμίσεων και θα ήθελα να πω ότι υπευρύθησαν 141 τροπολογίες από τα μέλη και ο εισηγητής ο κ. Χουντής έχει συντάξει κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χουντή, ο οποίος θα περιγράψει τη θέση του όσον αφορά τις τροπολογίες. Έχετε το λόγο κύριε Χουντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ τη Γραμματεία για την διαμόρφωση του προγράμματος, τη Γραμματεία της Επιτροπής μας, με σκοπό να γίνει δυνατή αυτή την ώρα η συζήτηση της έκθεσης. Ήταν μια δικιά μου παράκληση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την πρώτη συζήτηση που κάναμε για το σχέδιο έκθεσης για την ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας και αφού από τη συζήτηση φάνηκε ότι στα βασικά συμφωνούμε τουλάχιστον όσοι είχαν μιλήσει, όσοι και όσες είχαν μιλήσει και αφού συμφωνούμε και στο κρίσιμο θέμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση να δοθεί καθεστώς ε, υποένταξη μέλους στην Αλβανία ε, στα επιμέρους θέματα ή και γενικά κατατέθηκαν όπως είπε ο αγαπητός Πρόεδρος 141 τροπολογίες. Ε, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που κατέθεσαν αυτές τις τροπολογίες γιατί βοηθούν στην καλύτερη διαμόρφωση της έκθεσης. Για να μην τρώω πολύ χρόνο, ε, θέλω να σας πω ότι έγινε μια προσπάθεια να γίνει συνάντηση των Σάντοους, αλλά των σκιωδών εισηγητών, αλλά λόγω αντικειμενικής αδυναμίας από ό,τι ενημερώθηκα των ε, σκιωδών εισηγητών δεν έγινε δυνατή μια τέτοια συνάντηση. Ε, από τις τροπολογίες που κατετέθηκαν... Ε, ε, έχουν διαμορφωθεί οι, οι συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες έχετε μπροστά σας που μοιράστηκαν από ό,τι είδα και σήμερα νομίζω πρέπει να τις έχετε έγκαιρα θα τις έχετε πάρει σε αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες πήρα παρατηρήσεις γραπτές εκ μέρους του EPP από την κυρία Πακ και την ευχαριστώ γι' αυτό και επομένως μια σύντομη παρουσίαση στο που βρισκόμαστε σήμερα στις συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν σχέση με αυτόν τον διάλογο ας πούμε και τις παρατηρήσεις της κυρίας Πακ ε, κατά βάση. Δεν λέω ότι δεν ε, υπάρχουν και οι άλλες τροπολογίες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη αλλά για να προχωρήσουμε παραπέρα τα πράγματα. Ε, να πω ότι πριν πω επί της ουσίας, ότι μέχρι το απόγευμα 6 ώρα πρέπει να έχουμε καταλήξει να υπάρχουν περαιτέρω ας το πούμε τροπολογίες ή παρατηρήσεις ή συμφωνίες ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο να υπάρξει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και να πάμε μετά στην Ολομέλεια. Ε, τώρα, ε, ε, όσο αφορά την πρώτη τροπολογία δεν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις ε, Περιτώ να πω ότι εδώ ενσωματώνονται τροπολογίες που με διαφορετικές διατυπώσεις λένε το ίδιο πράγμα. Αυτό ισχύει για όλες τις τροπολογίες. Επομένως, αν κάποιος συνάδελφος δεν βλέπει την ακριβή έκφρασή του, δεν σημαίνει διαφωνία επί της ουσίας και επομένως δεν, ε, όπως άλλωστε έτσι γίνεται. Επομένως, στην πρώτη ε, συμβιβαστική τροπολογία δεν έχω κάποια παρατήρηση έτσι όπως την έχετε μπροστά σας και μπορεί να γίνει δεκτή, αυτό συμπεραίνω, εκτός αν υπάρξουν μέχρι το απόγευμα, άλλες παρατηρήσεις. Το ίδιο και με τη δεύτερη τροπολογία, τη συμβιβαστική επαναλαμβάνω, που καλύπτει τις συγκεκριμένες τροπολογίες που αναφέρονται μέσα στην παρένθεση. Η παρατήρησή μου εδώ είναι ότι στο τέλος, στην τελευταία παράγραφο της δεύτερης συμβιβαστικής τροπολογίας, στην 2α, στη δεύτερη σελίδα του εντύπου που έχετε μπροστά σας, όσο αφορά τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας για την Ευρώπη υπάρχει μια γλωσσική αλλαγή γιατί σύμφωνα με αυτό που προτείνει και η Κομισιόν και ισχύει δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις του οργανισμού για την Αλβανία υπάρχουν γενικές αρχές με τις οποίες καλείται να συμμορφωθεί και η Αλβανία. Αυτό εξυπηρετεί η γλωσσική διαφορά. Στην παρατήρηση στο τροπολογία αριθμό 3, τη συμβιβαστική πάλι, εδώ, αγαπητέ Πρόεδρε, μια πρότασή σας, μια λέξη σας σχετικά με το limited στην τροπολογία τι, τι προόδοι έχουν γίνει, θα έλεγα να τη, βγάζουμε, να τη βγάζαμε αυτή τη λέξη και να πούμε ότι έγιναν κάποιοι πρόοδοι αναγνωρίζοντας αυτό που λέει και η πρόοδος της Κομισιόν. Είναι φραστικό, έχει τη σημασία του και αυτό. Η πρόταση που κάνω είναι να πούμε έχουν γίνει κάποιοι πρόοδοι. Επίσης το στην ίδια συμβιβαστική τροπολογία στο 7α. Ε, εδώ βγάζουμε την πρόταση από την τροπολογία της κυρίας Κορνέλιασεν ε, διότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία από ούτε από την Κομισιόν που να στοιχειοθετούν ότι η εκτεταμένη διαφθορά στο δικαστικό σώμα και ότι εμποδίζεται η εφαρμογή των σχετικών νόμων για το τράφικινγκ ενώ κρατάμε το υπόλοιπο της ε, τροπολογίας. Να το ξαναπώ, δεν έχουμε στοιχεία ότι εμποδίζεται η εφαρμογή των νόμων για το τράφικινγκ, γι' αυτό κάνουμε την ε, αλλαγή αυτή. Όσο αφορά την τροπολογία 4, δεν έχω κάτι να πω, κάτι, δεν μου παρατηρήθηκε κάτι το συγκεκριμένο. Όσο αφορά την τροπολογία 5, από ό,τι είδα από τις προτάσεις, από την παρατήρηση της κυρίας Πακ, ε, δεν έχουμε συμφωνία σε αυτό το σημείο. Ε, εγώ επιμένω, είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και πάση περιπτώσει νομίζω ότι πρέπει να περιέχονται στην έκθεση και γενικώ, ε, για να μην τα αναφέρω και σε άλλες τροπολογίες, διότι εμφανίζονται και παρακάτω, οι παρατηρήσεις εκ μέρους του ΕΠΠ έχουν κυρίως να κάνουν με θέματα δικαιωμάτων εγώ νομίζω ότι πρέπει να μείνουν αυτά τα θέματα, μπορούμε να επιμείνουμε γενικώ. Γι' αυτό με βλέπετε να είμαι αντίθετο στο να φύγουν όπω προτείνει η κυρία Πακ, ε, το ΕΠΠ δεν γνωρίζω αν είναι συνολική πρόταση. Ε, επίσης, ε, στην ίδια ε, τροπολογία, στην τροπολογία 5, για τις μειονότητες, η τελική μου πρόταση είναι να αποφύγουμε να αναφερθούμε ειδικά στις δύο μειονότητες, Αρωμάνιανς και Ρωμά, διότι το γενικό πνεύμα και το νόημα και η αναφορά είναι για όλες τις μειονότητες. Άλλωστε η αναφορά στους Ρωμά υπάρχει και παρακάτω, θα ήταν πλεονασμός. Αυτή είναι η πρόταση στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή η τροποποίηση, η διαφοροποίηση, η αλλαγή στις, ε, ε, στην ε, τροπολογία τη συμβιβαστική που αναφέρομαι τώρα και είμαι στο σημείο 5. Και στο σημείο 6, στην τροπολογία 6, συγγνώμη, εκεί αλλάζουμε σε σχέση με την διατύπωση που έχετε μπροστά σας την ορολογία LGBT εδώ με το θέμα με τις ομάδες, με τη λέξη πρόσωπα γιατί νομίζουμε ότι δεν είναι καλό να κατηγοριοποιείς τους ανθρώπους λόγω σεξουαλικού προσδιορισμού με τη λέξη πρόσωπα και το νόημα της ε, τροπολογίας νομίζω ότι καλύπτεται αυτό το θέμα τη 15α στην επόμενη παράγραφο, παράγραφο υπήρξε μια παρατήρηση να βγει η λέξη, η έκφραση, το νόημα education, δηλαδή education σε σχέση με την εκπαίδευση, με το αιτιολογικό ότι τα κορίτσια είναι πιο πολλά από τα γόρια στην Αλβανία, έτσι, στα σχολεία και οι, δασκάλ, οι δασκάλες, οι δάσκαλοι θηλυκού γένους, περισσότερο από τους δασκάλους αρσενικού γένους, όμως η σημασία είναι γενικότερη και νομίζω ότι πρέπει να μείνει. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει επιμονή και θεωρείται τόσο σημαντικό, δεν νομίζω ότι ας το πούμε μπορούμε να, εδώ να, έχουμε, να συνεχιστεί η διαφωνία. Στην επόμενη παράγραφο 15β, ε, εδώ μ, φεύγει η φράση που αναφέρεται στη λειτουργία δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας και πάει πιο κάτω στο σημείο που καλωσορίζουμε τα όσα έχουν επιτευχθεί στο θέμα της προστασίας των θυμάτων της βίας, γιατί υπάρχει και λειτουργεί μια τέτοια, γραμμή, ε, μια τέτοια διαδικασία. Και εδώ δεν έχω κάποια παρατήρηση που να λέει το αντίθετο. Ε, πλησιάζουμε προς το τέλος για να μην τρώω πολύ χρόνο. Πάμε στην τροπολογία αριθμό 7. Ε, εδώ υπάρχει παρατήρηση από το EPP, από την κυρία Πακ, καλό είναι να μείνει η αρχική διατύπωση που είχε το κείμενο πριν μπούμε στη διαδικασία των τροπολογιών. Η πρόταση δική μου είναι να πάμε σε αυτή την τροπολογία γιατί περιέχει ε, ορισμένα πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα και για τα παιδιά, στοιχεία που σε μια συζήτηση με τη UNICEF μας ε, τα τεκμηρίωσαν και για τον εθνικό συνήγορο του πολίτη. Στην τροπολογία 8 δεν έχω κάτι μετά την τελική διατύπωση. Στην τροπολογία 9 είμαστε σύμφωνοι. Υπάρχει μια παρατήρηση στην τελευταία φράση σχετικά με την Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Υπάρχει μια ένσταση, αν κατάλαβα καλά, δεν την εστερνίζομαι και σύντομα λέω θα ήθελα να μείνει αυτή η τοποθέτηση. Υπάρχουν και σχετικές τροπολογίες ως προς αυτό. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε με την τελευταία συμβιβαστική τροπολογία και εδώ υπάρχει παρατήρηση ότι υπάρχει το θέμα της ανεργίας και μετά το συμπληρώνουμε και με προβλήματα άλλων κατηγοριών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συνόψη στη σχετική παράγραφο αυτών των θεμάτων σχετικά με τα πρόσωπα, με, τα παιδιά, συγγνώμη, με πρόσωπα με ανάγκες, ειδικές ανάγκες, ε, μειονοτικές ομάδες κτλ. Νομίζω ότι δίνει μια ενότητα σε αυτή την ε, συμβιβαστική παρατήρηση και η εισηγητική μου τοποθέτηση, ξεκινώντας τη συζήτησή μας λοιπόν, να ακούσω αν υπάρχει κάτι, νομίζω ότι πρέπει να μείνει. Ε, εδώ θέλω να σταματήσω κύριε Πρόεδρε, διότι καλό είναι να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, σκιώδης ή όποιος άλλος συνάδελφος έχει να παρατηρήσει αυτά, για να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε και πώς θα τελειώσουμε την προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστώ και πάλι όσους έχουν κάνει παρατηρήσεις και όσους θα λάβουν το λόγο για να συμπληρώσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντή. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές για τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Για το ΕΛΚ, η κυρία Πάκ είναι σκιώδης εισηγήτρια. Μου ζήτησε να παρουσιάσω τις τροπολογίες της και τα σχόλιά της. Θα καταλαβαίνετε συνάδελφοι πόσο δύσκολο είναι να αντικαθιστά κανείς την κυρία Ντόρις Πακ. Θα διαβάσω τα σχόλιά της. Παρόλο που ο κύριος εισηγητής ανέφερε αρκετές από τις τροπολογίες της και πάλι θα διαβάσω αυτά που μου έγραψε. Υποστηρίζουμε τις συμβαστικές 1, 2, 3, 4, 8 όσε προτάθησαν τη συμβαστική 5 είμαστε κατά της πρώτης παραγράφου διότι η χρήση των μειωνοτικών γλωσσών στην Αλβανία ήδη προβλέπεται στο Σύνταγμα καθώς και στην νομοθεσία. Άρα είμαστε υπέρ της δεύτερης παραγράφου της 14α όσον αφορά τις μειονοτικές ομάδες. Συμβαστική 6 προτιμούμε την αρχική παράγραφο, το πρωτότυπο η κυρία Πάκ υποστηρίζει γι' αυτό μόνο το πρώτο τμήμα της παραγράφου 15 ως έχει, ως ακολουθεί. Καλή για την αναγκαία πρόοδο στον τομέα των, ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των διαφόρων σεξουαλικών προτιμήσεων, δικαιωμάτων των παιδιών, των ευαλωτών ατόμων και των ατόμων με αναπηρίες. Η υπόλοιπη παράγραφος 15 μας βρίσκει αντιθέτους. Είμαστε υπέρ της παραγράφου 15 χωρίς τη λέξη εκπαίδευση, education, αυτό που είπε και ο κ. Συγητής, διότι ο αριθμός των γυναικών στα σχολεία στην Αλβανία είναι μεγαλύτερος από των ανδρών και επειδή οι γυναίκες δάσκαλοι είναι περισσότερες από τους άνδρες δασκάλους. Στην παράγραφο 15β είμαστε κατά αυτής. Συμβαστική 7 είμαστε κατά όλης της συμβαστικής τροπολογίας διότι πιστεύουμε ότι η αρχική παράγραφος 18 στο ψήφισμα είναι καλύτερη. Συμβιβαστική 9 μπορούμε να την αποδεχτούμε, αλλά είμαστε κατά της τελευταίας φράσης που καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των απαυλίτων και να δημιουργήσει μια υποδομή που λειτουργεί καλά όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Συμβαστική 10, είμαστε υπέρ της συμβαστικής από την αρχή μέχρι εκεί που λέει τους οικονομικά πιο αδύναμους πολίτες και εκείνους που έχουν περισσότερες ανάγκες. Είμαστε κατά του κομματιού που ακολουθεί που λέει συμπεριλαμβανομένων των ευαλώτων ατόμων σε, θέματα, σε υπηρεσίες υγείας και στέγασης αυτά θα έπρεπε να αφαιρεθούν από τη συμβιβαστική λύση διότι η παράγραφος εστιάζεται στο υψηλό επίπεδο της ανεργίας, υψηλό ποσοστό της ανεργίας. Όλες αυτές οι τροπολογίες αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και έχοντας ακούσει προσεκτικά τον κύριο Σιγητή είδα ότι δεν υπήρχε μεγάλη συμφωνία μεταξύ σχολείων του κυρίου Σιγητού και τα όσων λέει η κυρία Πακ, οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερες συζητήσεις για να επιτευχθεί μια ευρεία συμφωνία επί των συμβιβαστικών. Για το S&D Δίνω το λόγο στο διακεκριμένο συνάδελφο κύριο Ζάλα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της σοσιαλιστικής ομάδας συγχαίρω τον εισηγητή. Έξοχη η δουλειά που έκανε για το σχέδιο έκθεσης και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Η ομάδα μας υποστηρίζει όλες τις συμβαστικές τροπολογίες που μας προτείνει. Εν γέννη η έκθεση δίνει το σωστό πολιτικό τόνο, κυρίως συμβαστικές 1, 2, 3. Πρώτα απ' όλα αντικατοπτρίζεται ισχυρή υποστήριξη του Κοινοβουλίου για το να είναι υποψήφια χώρα η Αλβανία για προσχώρηση υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι βραχυπρόθεσμοι όροι προϋποθέσεις και ότι θα υπάρξει ε, υποστήριξη της συνεργασίας του Κοινοβούλου. Καθιστά καθαρό ότι είναι κρισίμου σημασία οι κοινοβουλευτικέ ε, εκλογές για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δοκιμαστεί η δημοκρατική οριμότητα της Αλβανίας. Η Αλβανία πέρα από αυτού έχει πολύ σοβαρές προκλήσεις να αντιμετωπίσει για να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενώσης, κυρίως για το κάτω δικαίου και για την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, στη διαφύλαξη ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά υπάρχει ένα γενικό πνεύμα ανοίγματο, υπάρχει πολιτική, έχει ανοίξει ένα πολιτική δυνατότητα για να προχωρήσει και να κάνει άλμα η Αλβανία για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους μήνες. Οι σημαστικές τροπολογίες ενισχύουν αυτό το μήνυμα της ευκαιρίας που δημιουργείται, αλλά αναφέρουν και τους όρους που θα πρέπει να πληρούνται για κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή και πλήρης έκθεση. Η ομάδα μας με χαρά μπορεί να ε, υποστηρίξει την έκθεση αυτή στην ψηφοφορία στην ΑΦΕ την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζάλα για τους πρασίνους. Η κυρία Κορνέλισεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χουντή για τη δουλειά που έκανε και άκουσε τις απόψεις. Χαιρόμαστε πολύ για τις συμβαστικές που προτείνει και πολλές ομάδες πιστεύω ότι συμφωνούν θα μπορεί να τύχει το κείμενο υποστήριξης ευρύτερης από πολλά κόμματα ε, για τη συμβαστική 2 Χαίρομαι για το κείμενο που βλέπω. Είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό κλίμα και η διακομματική συνεργασία να υπάρχουν. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που έχουμε όσον αφορά την Αλβανία και η ένα, είναι καλή, είναι σαφέστατο εκεί ότι υποστηρίζουμε την έκκληση ε, να γίνει η Αλβανία υποψήφια χώρα, αλλά πρέπει να πληρούνται πρώτα κάποια κριτήρια. Και δεν μπορούμε εκεί να είμαστε ελαστικοί όσον αφορά τα κριτήρια. Μας ικανοποιεί πολύ και η συμβαστική 6, όπου είναι πολύ σημαντικό το θέμα, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται. Μία ερώτηση που αφορά το ΕΛΚ περισσότερο. Ο κύριος Κούκαν, εκ μέρους της κυρίας Πακ, είπε ότι δεν θέλετε να υποστηρίξετε αναφορά της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για τη Διαχείριση των Αποβλήτων και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Διότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αλβανία. Υπάρχουν πολλά απόβλητα, τοξικά απόβλητα που εισάγονται. Τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Θα ήθελα να μου δοθεί κάποια απάντηση από πλευράς ΕΛΚ πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον από την Αλτε ή από το ECR. Οπότε θα δώσω το λόγο στους άλλους συναδέλφους που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο για αυτό το θέμα και αν επιτρέπετε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Νομίζω ότι ήταν καλή συζήτηση όσον αφορά την έκθεση για την Αλβανία που έγινε την προηγούμενη φορά και ελπίζω ότι αυτή η καλή συζήτηση για τις τροπολογίες θα συνεχιστεί και αυτό θα βοηθήσει τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της έκθεσης που πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι κάτι επικοδομητικό. Κάποια σχόλια έχω για κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνώ και εγώ με τη συμβαστική 1, 2, 3 και 4. Στη συμβαστική 3, κύριε Σιγητά, το αναφέρεται, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα άξιζε τον κόπο να συζητηθεί έτσι περαιτέρω το τι είδους πρόοδος ακριβώς έχει αντικειμενικά και δίκαια επιτευχθεί στην Αλβανία. Δεν προτείνω κάποια τελική λύση γι' αυτό, αν είναι πρόοδος ή περιορισμένη πρόοδος. Όσον αφορά τη συμβαστική 1, συμφωνώ, αλλά ολοκλήρωση, completion είναι η βασική ενα συμφωνω αλλα ολοκληρωση completion ειναι Η ολοκλήρωση της εκκρεμούσης εκθέσεως και η έγκριση και εφαρμογή adoption και implementation. Αυτή τη γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιούμε σε όλες τις παραγράφους στο, στην έκθεση. Συμβαστική δύο, συμφωνώ. Πράγματι συνεργασία μεταξύ της κυβερνούσης πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι κάτι που βελτιώνει το πολιτικό κλίμα, αποτελεί επανάληψη, αναφέρεται δύο φορές σε μία σύντομη παράγραφο. Συμφωνώ με αυτό, αλλά θα ήθελα να πω ότι εγώ ίδιος χρειάζομαι αποδείξεις, πραγματικές αποδείξεις να με βοηθήσουν να ξεπεράσω τους δισταγμούς που έχω, το στεπτικισμό μου, δηλαδή κατά πόσο πράγματι αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ε, Αλβανία. Το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής αυτής αναφέρεται στις εκλογές, αποδεκτό αυτό. Βέβαια θα είναι πολύ σημαντικό για την Αλβανία το πώς θα διεξαχθούν οι επικείμενες εκλογές, πώς θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, ποια συνέχεια θα δοθεί, τι θα ακολουθήσει τις εκλογές. Δύο δικές μου τροπολογίες θα ήθελα να τις διατηρήσω. Η τροπολογία 74 αναφέρεται στην έρευνα του γεγονότος της 23ης Ιανουαρίου. Είναι σημαντικό για την Αλβανία και για τους πολίτες της αυτά τα γεγονότα να ερευνηθούν κανονικά και ανεξάρτητα μέσω μιας και να ξεκινήσει μια αξιόπιστη νομική δικαστική διαδικασία. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα είναι κάτι καλό για την κοινωνία στην Αλβανία. Δεύτερον, έχουμε την τροπολογία 133 που υπέβαλα μετά από την έντονη κατάσταση όταν πρώην πολιτικοί φυλακισμένοι κάναν απεργία και δύο από αυτούς αυτοπυρπολήθηκαν. Ξέρω ότι άλλαξε η κατάσταση έκτοτε, αλλά θα ήθελα να παραμείνει η τροπολογία και αν είναι αναγκαίο θα υποβάλω προφορική τροπολογία για να αντικατοπτρίζεται αντικειμενικά και καλύτερα η παρούσα κατάσταση. Αυτά τα σχόλια έχω και θέλω να δω αν υπάρχει κάποιος άλλος. Ο κύριος Βιγγένιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαίρω τον εισηγητή για την έκθεση και τις συμβαστικέ τροπολογίες που ετοίμασε. Βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποιες από αυτές και ο σκιώδης εισηγητής των ε, σοσιαλιστών θα συμμετάσχει σε αυτό. Τι έχω να πω, ότι οι τροπολογίες μου κυρίως αυτές που αφορούν το πολιτικό κλίμα στην χώρα, αντικατοπτρίζονται σωστά στις τροπολογίες, τις συμβαστικές και είμαι ικανοποιημένο. Όμως, να πω κάτι, γιατί είναι καλή ευκαιρία αυτή. Να το συζητήσουμε. Να πω το εξή λοιπόν. Όσον αφορά το πολιτικό κλίμα, έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα. Και ένα από τα ζητήματα που θα έπρεπε να δημιουργούν ανησυχίες για το Κοινοβούλιο είναι ότι τρεις νομοθετικές πράξεις που θα πρέπει να εγκριθούν, ούτω ώστε η Αλβανία να ελπίζει να θεωρηθεί υποψήφια χώρα φαίνεται ότι δεν την χάνουν τις αναγκαίες υποστήριξης στο Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης επ' αυτών και επί άλλων ζητημάτων σχετικών. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρίες να καλέσω και αντιπολίτευση και κυβέρνηση να βρουν γρήγορα μια λύση στο ζήτημα. Διότι είναι δυνατός ένα συμβιβασμός, δεν είναι τόσο σοβαρά αυτά τα προβλήματα και δεν θα ήταν δίκιο να κατηγορούμε εδώ την αντιπολίτευση, να τη θεωρήσουμε ότι δεν θέλει να υποστηρίξει αυτά τα νομοσχέδια γιατί είναι και θέμα της κυβέρνησης. Και η κυβερνητική πλειοψηφία θα πρέπει να καταλάβει τη σημασία που έχουν αυτοί οι νόμοι και το βήμα που πρέπει να γίνει, ούτως ώστε ε, να κάνουν και τις αναγκαίες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Αν δεν υιοθετηθούν αυτά τα νομοσχέδια, δεν μπορεί να ελπίσει η χώρα να γίνει υποψήφια τώρα. Ίσως να μην το καταφέρουν αυτό, ακόμα και αν υιοθετηθούν αυτοί οι νόμοι, αλλά έχουν περισσότερες πιθανότητες. Υπάρχουν ήδη χώρες που διατείνονται ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υποψήφια χώρα μέχρι τις εκλογές του χρόνου αλλά το Κοινοβούλιο θα ήθελε να δει η επίτευξη προόδου του ταχύτερο δυνατόν, γιατί θεωρούμε ότι τη στιγμή που θα γίνει υποψήφια αυτή η χώρα, θα ενθαρρυνθεί περισσότερο να διεξαγάγει ελεύθερα και δίκαια τι επόμενε εκλογέ. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα, αν τη χορηγηθεί καθεστώ υποψήφια χώρα. Γι' αυτό και αντιπολίτευση και κυβέρνηση θα πρέπει να δείξουν ότι είναι αφοσιωμένοι προ τον ευρωπαϊκό στόχο και να κάνουν τι αναγκαίε υποχωρήσει. Αν δεν το δούμε αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι πραγματικά η χώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση πάνω σε αυτό το μονοπάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίγενίν, για τα εύστοχα αυτά σχόλιά σας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ζητάει το λόγο, αλλά πρωτού δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαραγκό από τη Γενική Διεύθυνση Διεύθυνσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στη διατύπωση αυτού του ψηφίσματος για την υποστήριξη που δίδεται στην πρόταση της Κομισιόν και την ανάλυση της Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι η Αλβανία έχουν κάνει, έχει κάνει σημαντική πρόοδο εφέτος, ιδίως στα πλαίσια της πολιτικής συμφωνίας του πρόσφατου Νοέμβρη τον προηγούμενο Νοέμβρη που έχει αρχίσει και η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και σε άλλους τομείς μεταρρύθμισης όπως αναφέρουμε στην έκθεση πρόοδου και στο έγγραφο στρατηγικής. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους φίλους της Αλβανίας, τους φίλους μας στην Αλβανία, ένα μήνυμα ότι τους ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν και σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Όπως ελέγχθη από πολλού ομιλητέ, το θέμα τη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι κεφαλαιόδε ναι. ώστε η Αλβανία να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε μια ενωμένη άποψη για τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να προστοκούμε περαιτέρω συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία. Αλλά όπως είπε και ο κ. Βίγκενεν, είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτική διαδικασία στην Αλβανία να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό χωρίς να βασίζεται μονάχα στην πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για ένα ή δύο θέματα που αναφερθήκαν, να τονίσω ότι για μας το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρθηκε προηγουμένως από την κυρία Κονέλσεν πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Φυσικά εσείς θα αποφασίσετε πώς θα διατυπώσετε το θέμα αυτό, αλλά είναι φυσικά πολύ σημαντικό να τονίσουμε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, όχι μόνο στο πλαίσιο των εισαγωγών, αλλά και για να εξασφαλιστεί μια σωστή λειτουργία της διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στις διμερείς επαφές μας με την Αλβανία και ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπιστεί και στην επόμενη φάση του προγράμματος αντικτύπου το οποίο ξεκινάει. Το δεύτερο αφορά τη δικαστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία είναι ένας χώρος όπου πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν. Εφέτος όμως έχουν ήδη γίνει σημαντικές πρόοδοι και μία από αυτές τις πρόοδους ήταν η μεταρρύθμιση των κανόνων για την ασυλία. Έρεται η ασυλία του δικαστικού τομέα και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστούν τα θέματα διαφθοράς μεταξύ των δικαστικών και άλλα τμήματα της νομοθεσίας έχουν μεταρρυθμιστεί, έχουν τροποποιηθεί. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους δικηγόρους για το ανώτατο συμβούλιο δικαστικών, πώς θα πρέπει να εκλέγεται κτλ. Γίνονται λοιπόν σημαντικές ενέργειες σε σχέση με τις πειθαρχικές διαδικασίες ε, από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν βέβαια, απλώς αναφέρουμε τα σημαντικότερα μεταξύ των οποίων και η νομοθεσία για το Ανώτατο Δικαστήριο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι στο δικαστικό τομέα η πρόοδος στην Αλβανία εφέτος ήταν κάπως μέτριοπαθής, όπως λέμε στην εκθεσή μας, αλλά όχι περιορισμένη. Αυτή είναι φυσικά η δική μας κρίση και σε εσάς συναπόκειται πώς θα αξιολογήσετε την πρόοδο η οποία έχει γίνει από την Αλβανία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαραγκό. Κύριε Μαραγιά και δίνω το λόγο στον κύριο Χούντι για να κλείσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλους και όλες που πήραν το λόγο, πήρατε το λόγο και ε, αναφερθήκατε στις συγκεκριμένες τροπολογίες. Πριν πω στο πώς ε, βλέπω τις παρατηρήσεις που κάνατε, ε, θέλω να πω ότι πράγματι ενώ η έκθεσή μας δεν πρέπει να είναι πολύ παρεμβατική, δασκαλίστικη θα έλεγε κανείς, θα πρέπει να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ανησυχία μας για τη σταθεροποίηση του πολιτικού κλίματος και του διαλόγου, διότι όπως είχα πει και στην παρουσίαση στην, αρχική, στην προηγούμενη συζήτηση, δεν έχει σταθεροποιηθεί πλήρως για να πούμε ότι θα λυθούν σίγουρα τα προβλήματα αν δεν καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια. Και εδώ νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι να εκφράζεται αυτή η απαιτητικότητα των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρωθούν χωρίς καμία επανάπαυση από την πλευρά των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών της Αλβανίας. Τώρα, στα επιμέρους, στα θέματα των τροπολογιών, ε, θα ήθελα να σας πω ότι αμέσως μόλις τελειώσει η συνεδρίαση θα, θα στείλω σε όλους τους κοιόδης συζητητές τις μικρές τεχνικές ή γλωσσικές αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκα προφορικά, ούτως ώστε εγκαίρως να τις έχουν μπροστά τους γιατί πρέπει αυτή η συζήτηση να τελειώσει μέχρι τις 6 για να μπορέσουμε να, όπως με έχει ενημερώσει η Γραμματεία, για να μπορέσουμε να γίνει και η τελική voting list. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν τροπολογίες τις οποίες αναφέρθηκαν συνάδελφοι, κυρίως ο κύριος Κούκαν, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά εγώ στη Βόλ την λίστη, η δική μου γνώμη είναι να ψηφιστούν. Και αναφέρομαι κύριε Κούκαν ε, σε δύο που αναφερθήκατε πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή στην τροπολογία 74 είμαι θετικός, να γίνει έρευνα για τα γεγονότα του Γενάρη κτλ. Είμαι θετικός, ναι. Και επίσης και στην τροπολογία σας με τον αριθμό 133 για τα δικαιώματα των πρώην πολιτικών κρατουμένων. Είμαι θετικός. Στη voting list θα προτείνω να το ψηφίσουμε απλώς δεν καλύπτονται με, τα, με τις συμβιβαστικές προτάσεις ε, που κάνουμε. Τώρα, σε σχέση με τις ε, συμβιβαστικές προτάσεις, ε, κύριε Κούκαν, η πρώτη συμβιβαστική πρόταση την ενίσχυση με το γεγονός της υιοθέτησης εφαρμογής της, ε, που λέτε, να τα συμπληρώσουμε αυτό υιοθέτησε εφαρμογή. Αν θέλετε να μου στείλετε και την ακριβή διατύπωση, το βρίσκω σωστό και το αποδέχομαι να μπει. Είναι σωστό αυτό. Ε, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ με τη συζήτηση που κάναμε. Επίσης ε, δεν επιμένω για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Δεν επιμένω στο θέμα της education στην, ε, στο 6 εκεί που δεν θέλετε να μπει αυτό το θέμα, δεν, δεν επιμένω σε αυτό το συζήτημα. Και επίσης και στο 10 θα μπορούσε η τελευταία παράγραφος να φύγει αφού το ξανακοιτάξουμε αν αναφέρονται σε άλλα σημεία αυτά τα θέματα. Τώρα, ε, υπάρχει η τροπολογία 3 για το... Είναι και ουσία συζήτηση τι, τι, τι πρόοδοι έχουν γίνει στην Αλβανία και πώς θα τις χαρακτηρίσουμε. Και εδώ πάλι έχουμε όλη την αίσθηση ότι έχουν γίνει κάποιοι πρόοδοι, έχουν γίνει ορισμένες πρόοδοι, αλλά περιμένουμε περισσότερα. Δεν θα, δεν θα, δεν θα επιμείνω να είναι η δική μου ορολογία η καλύτερη, αν το limited σας εκφράζει καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι είναι περιορισμένες κάποιες που πρέπει να δώσουμε όθηση. Αν επιμένετε δεν έχω καμία αντίρρηση τελικά ότι μπορεί να γίνει αυτά τα θέματα. Ναι, ε, επίσης ε, δεν μπόρεσα να συγκρατήσω κύριε Κούκαν τι ακριβώς θέλετε ακριβώς το 2 να μπει. Δεν κατάλαβα το τέτοιο. Αν θέλετε στείλτε μου κάτι συγκεκριμένο έτσι για να με βοηθήσει για την τελική διατύπωση. Τώρα από τις, ε, ευχαριστώ τις, τους άλλους κοιόδης συγητές για τα σχόλιά τους και για τις υπογραμμίσεις τους. Στα σημεία που δεν αναφέρθηκα ότι, εν πάση περιπτώσει, μετά τη συζήτηση θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν οι διατυπώσεις, ε, σημαίνει ότι επιμένω να μείνουν. Και αναφέρομαι και στο, ε, στην ε, συμβιβαστική εννιά και για το Εθνικό Σχέδιο για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων και ότι αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια ένσταση από την πλευρά του, του Λαϊκού Κόμματος και κυρίως της κυρίας Πάκο, όπως τουλάχιστον με έχει πληροφορήσει και όπως μας είπε ο κύριος Κούκαν. Α, δεν νομίζω ότι ξεχνώ κάτι. Επομένως, ε, είναι φανερό ότι μέχρι το, τις 6 περιμένω τις παρατηρήσεις. Είναι φανερό ότι σε ορισμένες συμβιβαστικές προτάσεις, από ό,τι φαίνεται τις περισσότερες, θα είμαστε όλοι μαζί. Σε ορισμένες που, αν υπάρχει επιμονή, είπα εγώ πώς το βλέπω τελικά, θα πάμε με διαφορετικό τρόπο. Ναι, Αυτά ήθελα να πω πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σίγητα. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτησή μας για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η ψηφοφορία για το ψήφισμα αυτό θα λάβει χώρα στις 27 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. 22, 22, συγγνώμη, 22 στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τώρα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος ώρα Αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να καλωσορίσω θερμά εκ μέρου του κ. Χέλμαρτ Μπροκ, του Πρόεδρου, ο οποίο δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τον πρέσβη Ραβ, που είναι επικεφαλή τη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Σκόπια. Θα συζητήσουμε μαζί την κατάσταση στην τέτοια Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και μάλιστα θα επικεντρωθούμε ιδίως την προετοιμασία της προσένταξη. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πριν αναλάβει τα καθήκοντά του που όταν έλαβε τον Μάρτιο του 2012 ε, ακολούθησε μια εξαιρετική καριέρα διπλωμάτη και μεταξύ άλλων ήταν πρέσβη στην ε, Τουρκία. Αγαπητέ κύριε πρέσβη, γνωρίζετε ότι στηρίζουμε τις ε, διαπραγματεύσεις προς ένταξη της τέσσερις γιουσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και πιστεύουμε ότι διμερεί θέματα δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο σε αυτό. Στηρίζουμε επίσης ε, διαπραγματεύσεις για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση όσον αφορά το όνομα, θέμα που υπάρχει με την Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποιες είναι οι δικές σας οι απόψεις για τις προοπτικές μιας τέτοιας συμφωνίας. Όμως πρέπει να γίνουν και περισσότερα πράγματα από πλευρά τη χώρα όσον αφορά τι μεταρρυθμίσει. Θέλω λοιπόν να ξέρω πώ προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις εκεί σε τομεί όπω είναι ο δικαστικό τομέα, η καταπολέμηση τη διαφθοράς, η ελευθερία των μέσων ενημέρωση, ο διάλογο υψηλού επίπεδου ε, για την ε, προσχώρηση σίγουρα αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε. Πριν ε, όμως μπούμε στη συζήτηση, θα ήθελα προηγουμένως ο κύριος Χατζημαρκάκης να πάρει το λόγο, μια που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας ε, για ε, τις σχέσεις με τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να δώσω τις καλύτερες μου ευχές στον νέο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Όραμ. Θα διαδραματίσει φυσικά ένα ιδιαίτερο ρόλο το γνωρίζει και ο ίδιος και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε επιπλέον, επιτέλους ένα μόνιμο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια. Η τελευταία συνάντηση της ε, Σομπράνια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έλαβε χώρα στα Σκόπια τον Οκτώβριο όπως ε, προβλέπετε, λόγω της ασθένειας του συμπροέδρου μου και έχει μεταφερθεί στα μέσα Φεβρουαρίου. Αυτό είναι κρίμα γιατί είχαμε θεωρήσει ότι μπορούσαμε να διαδραματίσουμε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Αλλά φυσικά είναι σημαντική και η ευκαιρία αυτή που έχουμε τώρα κύριε Όραμ να ανταλλάξουμε απόψη μαζί σας. Η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει ξεκινήσει τις ε, μεταρρυθμίσεις της ήδη από τον προηγούμενο χρόνο και έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να μπορέσει να καλύψει τις προϋποθέσεις για ένταξη, παραμένουν τα θέματα της αντιμετωπίσης της ε, ε, διαφθοράς, της δικαστικής μεταρρύθμισης, της ε, μεταρρύθμισης του διοικητικού μηχανισμού. Πιστεύω ότι και από τις δύο πλευρές. Μπορεί να υπάρξει μια πρόοδος και στα πολιτικά θέματα. Υπήρξε όμως ένα σημαντικό πρόβλημα με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και πριν από ένα χρόνο υπήρξε μια σημαντική πρόοδος με την συζήτηση γύρω από μια στρογγυλή τράπεζα για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία του διαλόγου υψηλής, ε, υψηλού επίπεδου και με τη συμμετοχή του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Αρίφη και σίγουρα έχει συμβάλει αυτός ο διάλογος για την πρόθεση των θεμάτων αυτών. Φυσικά δεν αποτελεί υποκατάστατο για διάλογο για τα θέματα όπως ανέφερε και ο πρόεδρος μας του ονόματος της χώρας αυτής. Έχει ανοίξει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας, έχει δημιουργηθεί μια πρόοδος με μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των κυρίων Ποπόφσκι και Αβραμόπουλου, των Υπουργών Εξωτερικών. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία να ευδοκιμήσει αυτή η πρωτοβουλία. Υπάρχουν πολλά θετικά, θετικές ενδείξεις αλλά και αντικές ενδείξεις. Παρακολουθούμε μια δύσκολη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί και μεταξύ της ε, Σόφιας και των Σκοπιών που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο αλλά η χώρα μου, επίσης η Γερμανία, ε, βρίσκει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα για το θέμα των προξενικών θεωρήσεων και ζητά να επανεξεταστεί το θέμα αυτό. Τούτων λεχθέντων, εγώ θέλω να σας καλωσορίσω στον νέο ρόλο σας και θα ήθελα να σας τονίσω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθεί η χώρα αυτή το ταχύτερο δυνατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρέσβη. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ για ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή σας. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους σας για τη δουλειά που κάνετε εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και τη δουλειά που έκανε ο κύριος Ρίτσαρτ Χάουετ για το ΦΥΡΟΜ και τη δουλειά που κάνει. Θα ήθελα να εστιαστώ επί τριών ζητημάτων Πρώτα απ' όλα η μεταρρυθμιστική διαδικασία στη χώρα, δεύτερον πολιτικές εξελίξεις από όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου στη χώρα 1η ε, Μαρτίου και τέλος ε, κάποιες προκλήσεις μελλοντικέ. Αν αναφερθούμε στη μεταρρυθμιστική διαδικασία θα πρέπει να μιλήσουμε και για διάλογο για την ένταξη ψηλού επίπεδου που ξεκίνησε το Μάρτιο όταν ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση ο κ. Φούλε ήρθε στα Σκόπια και ξεκίνησε το διάλογο έδωσε εντελώς νέο δυναμισμό στις σχέσεις μεταξύ Σκοπίων ε, και, της και Βρυξελών, διότι πριν από αυτό δεν ήταν τόσο καλές οι σχέσεις. Αυτός ο διάλογος και η πρωτοβουλία ε, θεωρήθηκαν πολύ θετικά πράγματα στη χώρα και στην κοινωνία. Όλοι ήταν πολύ θετική η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, η κοινωνία των πολιτών. Ο κόσμος στους δρόμους μιλούσε για τον διάλογο υψηλού επίπεδου για την ένταξη. Και αυτό με εξέπληξε. Πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα συμφωνήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κυβερνήσεως και ήταν το πρόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ετέθη. Τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην έκθεση προόδου ε, ήταν επικρίσεις όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης στο κράτος δικαίου, δημόσια δίκη, αυτά τα προβληματικά σημεία, μεταρρύθμιση των, ε, όσον αφορά τις εκλογές και κίνηση προς την οικονομία της αγοράς. Ε, πολλοί στόχοι τέθησαν και ήταν πολύ δύσκολο να συμφωνηθούν επί χάρτου, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστούν από πλευρά κυβερνήσεως οι στόχοι. Είδαμε λοιπόν ότι όμως ήθελε διακαώς να εφαρμόσει του στόχου η κυβέρνηση αυτού που συμφωνηθεί και δεσμεύτηκε ο κύριο ο ε, και ο, κύριο κύριος ο αντιπρόεδρο ο Επίτροπος Φούλελ πήγε στη χώρα όσον αφορά το διάλογο αυτό υψηλού επίπεδου Μάρτιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Τρεις φορές ήρθε στη χώρα και η επόμενη επισκεφτή του είχε σχεδιαστεί για τον Ιανουάριο. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποια επιτεύγματα του διαλόγου υψηλού επίπεδου για την προσχώρηση. Η Συμφωνία Πλαισίου της Αχρίδας, ε, ε, η αποτίμηση που έγινε αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε η εργασία από την κυβέρνηση το 2001 ε, υπήρχαν εθνοτικέ συγκρούσει στη χώρα και υπεγράφει στο τέλο αυτή η συμφωνία πλαίσια από πολιτικού πολιτικούς και αυτή η συμφωνία που στηρίχθηκε ένθερμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη διεθνή κοινότητα. Όλοι στη χώρα τώρα κατανοούν πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία, Όμω, διαφορετικέ εθνοτικέ ε, κοινότητε ε, ερμηνεύουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικότατο ο συνασπισμό από Σλαβομακεδόνες και Αλβανούς αυτός ο συνασπισμός, ο κυβερνητικός να μπορεί να συμφωνήσει βλέποντας τι έγινε τα περασμένα δέκα χρόνια, τι ακριβώς έγινε και πώς εφαρμόζεται μέχρι τώρα αυτή η συμφωνία που επετέχθη. Είναι μια καλή βάση για περαιτέρω πρόοδο ε, για να δούμε στο μέλλον πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία πλαίσιο της Αχρίδας. Ε, δεύτερον, η εκλογική μεταρρύθμιση ο νέος εκλογικός νόμος εθετήθηκε πρόσφατα. Το 2011 έγιναν κοινοβουλευτικές εκλογές και για πρώτη φορά ε, διεξήχθησαν καλά και δεν υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά τις εκλογές. Ο ΑΣΕ ε, ήταν, ε, είχε στείλει παρατηρητές ε, στην, στις εκλογές και δόθηκαν κάποιες στάσεις από τους παρατηρητές όπως και για οποιοδήποτε άλλη χώρα, ώστε και τελικά ενσωματώθηκαν στον εκλογικό νόμο οι παρατηρήσεις. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση να εφαρμόσει σωστά το νόμο που ψηφίστηκε. Τρίτο επίτευγμα, το κράτος ε, δικαίου το Μάρτιο έγινε διαδικασία εξέταση των κεφαλαίων 23 και 24. Έγινε συζήτηση με το Μαυροβούνιο και προσεκλήθηκε η χώρα αυτή ως παρατηρητής. Ο, ο νόμος για τα δικαστήρια είναι στο Κοινοβούλιο η συζήτηση πιθανότατα θα αρχίσει το τέλος αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη εβδομάδα. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωση είναι από το πλέον ορατό ζήτημα. Ένα από τα βασικά θέματα του διαλόγου υψηλού επίπεδου, ενταξιακού διαλόγου, ο νόμος για την απο... Ε, επίσης και για την αποποινικοποίηση της, ε, της δυσφήμισης ε, είναι κάτι που ίσως και δεν έχουμε και σε κάποιες χώρες. Ε, σε κάποιες χώρες είναι αυτή η, η συκοφαντία, η συκοφάντηση είναι ποινικό αδίκημα. Ε, η Ένωση Δημοσιογράφων μας είπε ότι πραγματικά προωθείται αυτό το νομοσχέδιο στη χώρα και είναι πολύ θετικό. Εκπρόσωπος της σε έκανε κάποια δήλωση και καλωσόρισε αυτό το νόμο που πέρασε στη χώρα. Και κάτι άλλο όσον αφορά την ευθεία των μέσων ενημέρωσης, και είναι σημαντικό να αναφερθεί εδώ, είναι η απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εκπομπών Ραδιοτηλεοπτικό ε, ε, για τη σύγκρουση συμφερόντων ώστε να μην υπάρχει ε, πρόβλημα όσον αφορά την διοκτησία κάποιων ΜΜΕ. Κατά πολέμηση διαφθορά, να υπάρχουν πολλέ προκλήσει όπω αναφέρατε, αλλά το βασικό είναι ότι η νομοθεσία για τη σύγκρουση των συμφερόντων δυνάμωσε, δυναμώθηκε. Και η ενίσχυση τη οικονομία τη αγορά, η κυβέρνηση των Σκοπίων πιστεύει ότι η χώρα είναι έτοιμη για το καθεστώς μιας λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς. Στον ενταξιακό διάλογο ψηλού επίπεδου δημιουργήθηκε και άλλος διάλογος μεταξύ των φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με το θέμα και της κυβερνήσεως, ούτως ώστε οι διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπιστούν και βασικό πρόβλημα είναι η αγορά εργασίας. Βασικό θέμα, η κατάσταση αγορά-εργασία στη χώρα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου ενταξιακού διαλόγου υψηλού επίπεδου το Σεπτέμβριο, στο έγγραφο συμπερασμάτων που συμφώνησαν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καλέ γειτονικέ σχέσει ήταν θέμα που αναφέρθηκε, που είναι σημαντικότατο βήμα. Τώρα, βλέποντα τι έγινε του περασμένου μήνε, εγώ θα έλεγα ότι πολλά έγιναν όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη σημασία που έχει η διαφάνεια και η συμπερίληψη όλων. Και θα έλεγα ότι ο βαθμό συμπερίληψη όλων των φορέων και η διαφάνεια ήταν όλα στοιχεία που ενισχύθηκαν αυτού του μήνε γιατί αρκετέ ομάδε εργασία δημιουργήθηκαν. Υπήρχαν εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών, η αντιπολίτευση εκλήθη επίση και συζητήθηκαν οι διάφορε τροποποίησεις των νόμων. Σήμερα πάνω από 70% των ελόγω στόχων που είχαν συμφωνηθεί έχουν εν μέρη ή πλήρω ε, επιτευχθεί αλλά δεν έχουν γίνει τα πάντα, αλλά συνεχίζεται αυτό ο ενταξιακός διάλογος υψηλού επίπεδου. Εδόθηκε σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσει με τη χώρα και πιστεύω ότι ο ενταξιακό διάλογο υψηλού επίπεδου έδωσε άλλο ένα επιχείρημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε αυτή τη σύσταση. Τώρα ερχόμενο στι πολιτικέ εξελίξει, το 2011-2012 πολλά γεγονότα έγιναν ε, κυρίως αθλητικές εκδηλώσεις πολύ συχνά ε, θεωρήθηκαν ότι ήταν προβλήματα εθνοτικά. Δύο μέρες πριν ξεκινήσω τη δουλειά μου στα Σκόπια έγινε επεισόδιο στο Κόστοβαρ όπου αστυνομικοί εκτός υπηρεσίες Σλαβομακεδόνες διαφώνησαν με γείτονες για θέση στάθμευσης ε, και αποτέλεσμα δύο νεκροί έγινε πρόβλημα εθνοτικό από τα μέσα ενημέρωσης και κάποια πολιτικά κόμματα θέλησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το επεισόδιο. Σοβαρό γεγονός έγινε στις 12 Απριλίου όταν πέντε άντρες πυροβολήθηκαν, σκοτώθηκαν στα βόρεια ε, των Σκοπίων κοντά στη λίμνη Σμισκόφσκη και αρχές Μαΐου έγινε επιχείρηση αστυνομική και συνελήφθησαν διάφοροι ύποπτοι του Υπουργείου Εσωτερικών ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν θρησκευ φανατικοί εξτρεμιστές που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Αυτό δημιούργησε πολλές παρεξηγήσεις κυρίως μεταξύ των ε, αλβανιοφωνών κοινοτήτων ε, και το αποτέλεσμα ήταν ε, μεγάλες διαμαρτυρίες στον δρόμο. Η Ισλαμική κοινωνία ε, είπε, η Ισλαμική κοινότητα ότι αυτό ήταν προσβολή για όλους τους μουσουλμάνους στη χώρα και οι εθνοτικοί Αλβανοί θεώρησαν ότι όλα αυτά είναι σκηνοθετημένα είναι πολύ, ήταν πιο περίπλοκα αυτά τα επεισόδια που συνέβησαν από άλλα και πριν το επεισόδιο Σμιλκόφσκι οι, οι εταίροι της κυβέρνησης πάντα κατάφερναν να δώσουν ενωτικά μηνύματα προς το κοινό μετά και ήταν κοινά μηνύματα μετά τα διάφορα κόμματα ε, της ε, κυβέρνησης άρχισαν να, να δίνουν διαφορετικά μηνύματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν ε, κάποιες ανακοινώσεις, μιλήσαν πολιτικούς ηγέτες, ε, παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα, συντονίσαμε ε, με τη ΣΥΠΑ, τις δηλώσεις με τον ΝΑΤΟ και με τον ΟΑΣΕ. και τα μηνύματά μας ήταν ότι βεβαίως το δικαίωμα του να μπορούν να συγκεντρώνονται οι άνθρωποι έπρεπε να διατηρηθεί. Αλλά δεν ήταν ώρα για ταραχές, ήταν σημαντικό να επικρατεί ηρεμία και υπευθυνότητα. Λοιπόν, ε, σήμερα έξι άτομα αντιμετώπισαν την κατηγορία της τρομοκρατίας και είναι πολύ σημαντικό οι δίκες να διεξαχθούν σωστά, ούτω ώστε να γίνει σωστός χειρισμός της πολιτικής καταστάσεως στη χώρα. Ε, είναι καλό ότι υποσχέθηκε ο Ασένα ε, να στείλει παρατηρητές στη δίκη και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενώσης στη χώρα συνεργαστεί με το φορέα αυτό. Μετά από το γεγονός του Σμιλκόφσκι, και μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ η υποστήριξη στο, ε, μειώθηκε όσον αφορά το, τους εθνοτικούς Αλβανούς στην κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο στο Υπουργείο Άμυνα από του από τους μέλη του Συνασπισμού των Εθνικών Αλβανών ε, κατέθεσαν στεφάνι στο νεκροταφείο, στην τελετή, οι Σλαβομακεδόνες το θεώρησαν σαν πρόκληση και υπέβαλαν σχετικό ψήφισμα στο Κοινοβούλιο. Υπήρχε ο νόμος από το 2002 που έδινε δικαίωμα στα θύματα των δυνάμεων ασφαλείας στη χώρα. Το νέο νομοσχέδιο θέλει να ωφελήσει περισσότερο αυτούς που εργάζονται στις δυνάμεις ασφαλείας. Όμως αυτό είναι απαράδεκτο για τους εθνοτικούς Αλβανούς που είναι στην κυβέρνηση γιατί θέλουν να συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι στο νομοσχέδιο. Αν εθετηθεί ο νόμος ως υπευλήθη στο Κοινοβούλιο θα είναι αδύνατον ε, τα μέλη του συνασπισμού Εθνοτική Αλβανοί να συνεχίσουν να παραμένουν στον συνασπισμό. Ο Πρωθυπουργό είπε δημόσια ότι αντιμετωπίζει κρίση η κυβέρνηση και θα γίνουν πρόωρα εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από όλου του εταίρους να δείξουν υπευθυνότητα και να επιδείξουν ηρεμία. Το νομοσχέδιο συζητείται στο Κοινοβούλιο και δύο κόμματα αλβανόφανα επέβαλαν πάνω από 1.500 τροπολογίε όσον αφορά το νομοσχέδιο. Θα συζητηθεί φαντάζομαι το νομοσχέδιο επί μακρόν. Υπάρχει εντύπωση ότι τα μέλη του συνασπισμού φαίνεται ότι συμφωνούν να διαφωνήσουν. Ερχόμενος τώρα στις διεθνείς σχέσεις Αρκετά βήματα έγιναν και αν μιλάμε για διεθνείς σχέσεις θα υπενθυμίζουμε εκεί και τις καλές γειτονικές σχέσεις. Δύο από τα κράτη-μέλη μας είναι γείτονες της εν λόγω χώρας και θα πρέπει οι ανησυχίες τους να γίνουν σεβαστές. Στις 5 Νοεμβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών και έστειλε μία επιστολή στον Έλληνα ομόλογό του απαντώντας στο, στο υπόμνημα συνεννόησης που απεστάλλει από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Στις 21 Οκτωβρίου ο Υπουργός Ποπός και έστειλε επιστολή στον Βούλγαρο ομολογό του προτείνοντας αρκετά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις διμερείς ε, σχέσεις. Στις 26 και 27 Οκτωβρίου ο Σέρβος Πρόεδρος επεσκέφθη τη χώρα ε, για να εορταστούν τα 100 χρόνια από τη μάχη του Κομάνοβο. Αυτή η μάχη είναι άκρος επίμαχη για τις αρχές των Σκοπίων. Ο πρόεδρος Ιβανόφ γι' αυτό δεν συμμετείχε στις εκδηλώσεις, αλλά οι αρχές των Σκοπίων δεν δημιουργούσαν πρόβλημα για τους Σέρβους όσον αφορά την τελετή. Αυτό το μήνα, ο ορτασμός των Κάποιο αλβανικό εορτασμό θα γίνει και ο πρόεδρο Γκουρέσκι θα πάει στα Τύρανα για τον εορτασμό και στι δημόσιε παρουσιάσει του ο πρόεδρο Γκουρέσκι ε, μίλησε αλβανικά. Εν κατακλείδη, υπάρχουν αρκετές εντάσεις, αλλά σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση μπορεί να τις αντιμετωπίσει τις εντάσεις και η κυβέρνηση είναι σταθερή. Όσον αφορά τις καλές γειτονικές σχέσεις, η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει πάρει πολύ σοβαρά το ζήτημα και προσπαθεί να βρει δυνατότητες για να προχωρήσει. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια προβλήματα, κάποιες προκλήσεις μάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις για τη χώρα αυτή και βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν στη χώρα η οποία είναι στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα αναφέρω πέντε τέτοιες προκλήσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι μετά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα προσθέσετε και άλλες και ίσως να δώσετε κάποιες ιδέες για την αντιμετώπιση τους. Λοιπόν, η πρώτη πρόκληση είναι η δίκη Σμιλκόφσκη. Όπως σας ανέφερα, είναι άκρος πολιτικής φύσεως αυτό το θέμα και διάφορες εθνοτικές ομάδες καταλαβαίνουν διαφορετικό τρόπο τη δίκη, γι' αυτό είναι σημαντικότατο η δίκη να διεξαχθεί πολύ σωστά και να υπάρχει από τον ΑΣΕ εκ του σύνεγγης παρατήρηση. Τοπικές εκλογές θα λάβουν χώρα τον Μάρτιο, δημοτικές εκλογές, και σίγουρα οι πολίτες στεστούν επί πολιτικών θεμάτων τοπικών στη χώρα, αλλά θα υπάρξουν ίσως και πειρασμοί να χρησιμοποιηθούν και διάφορα εθνοτικά ζητήματα στην προεκλογική εκστρατεία, οπότε κάθε προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί ούτως ώστε να ακολουθηθούν διεθνείς προδιαγραφές και νομίζω ότι η υιοθέτηση προσφάτως του εκλογικού νόμου είναι κάτι επικοδομητικό, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας εκλογικός νόμος πλήρως. Τρίτον, η εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας, που είναι, βασι... είναι κλειδί για τη σταθερότητα στην ε, χώρα, ανέφερα ήδη ότι η κυβέρνηση μπόρεσε να δει τι έγινε στο παρελθόν, να πετύχει συνένεση, ε, οι Σλαβομακεδόνες και οι Εθνοτικοί Αλβανοί να καταλάβουν με τον ίδιο τρόπο τι συνέβη τελευταία δεκαετία και αυτό αποτελεί πολύ καλή βάση για να προσβλέπουν προς το μέλλον και να έχουν ίδια αντίληψη για το μέλλον. Τέταρτον, μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να διατηρηθεί η ορμή τη μεταρρύθμιση και ο ενταξιακό διάλογο υψηλό επίπεδο αποτελεί άριστη βάση για κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρο ότι η κυβέρνηση θα δώσει συνέχεια στην προσπάθεια και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι και δικό τους. Βελτίωση της ορθής διακυβέρνησης προχωρά χέρι με χέρι με τους όρους για τις ξένες άμεσες επενδύσεις που είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και πέμπτον διατήρηση των προπτικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή είναι η ιδέα που ενώνει όλες τις κοινότητες της χώρας υπάρχει εθνική συνένεση για να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και μαζί με τη Συμφωνία Πλαίσιο της Οχρίδας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να συνεννοηθούν οι εθνοτικές κοινότητες χώρας και να κινηθούν με ειρηνικό τρόπο προς το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη για την πλήρη και λεπτομερή σας παρουσίαση και πολύ συγκεκριμένη θίξατε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική κατάσταση της ΦΥΡΟΜ. Τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Βίγκιανίν, ο οποίος θα μιλήσει εκ μέρους του μόνιμου συγκεκριτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΦΥΡΟΜ, του κύριο Ρίτσαρτ Χόβιτ, ο οποίος ε, ο ίδιος ε, πήρε την πρωτοβουλία για αυτή τη συνάντηση, αλλά δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, επειδή είναι σε αποστολή στη Σιέρα Λεόνε. Παρακαλώ, κύριε Βίγκιανίν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Ωρευ, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Το ότι ο κύριος Χόβουτ δεν είναι εδώ δεν σημαίνει ότι θα ήθελε να αποφύγει αυτή τη συνάντηση. Καθ' είναι παρατηρητής μας στις εκλογές εκεί. Γι' αυτό λείπει. Λοιπόν, εκ μέρους του κύριου Χόβουτ θέλω να σας πω ότι ανέλαβε πολύ σοβαρά τα καθήκοντά του. Έχει πάει στην Μακεδονία ολομιλητής τέσσερις φορές ε, ε, φέτο, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η τελευταία φορά, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, με υπουργού, με την αντιπολίτευση, με την κοινωνία των πολιτών και με τον κύριο Όραφ βέβαια. Και ένα από τα θέματα τα οποία θα ήθελε εδώ να μεταφέρει είναι ότι πρέπει να δούμε περισσότερο τις ευκαιρίες που υπάρχουν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει, να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών που είναι ένα από τα δύναμα σημεία από ό,τι φαίνεται σήμερα στη Μακεδονία. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σας μεταφέρω προς τον κύριο Όραφ εκ μέρους του Κοινοβουλίου και εκ μέρους του ίδιου του κύριου Χόβιτ είναι ότι η θέση του Κοινοβουλίου ήταν μια θέση αρχή τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει προκειμένου να υποστηρίξουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, προσχώρησης πιστεύουμε ότι τέτοιες διαπραγματεύσεις θα αποτελέσουν και όθηση και κίνητρο για τη χώρα να προχωρήσει σε αλλαγές. Είναι επίσης πολύ αισιόδοξο όσον αφορά ε, τον ε, διάλογο υψηλού επίπεδου που όντως έδωσε όθηση σε μεταρρυθμίσεις στη χώρα με αυτά αποτελέσματα. Όμως, αυτός ο διάλογος ε, προσχώρησης υψηλού επίπεδου πρέπει να δώσει όθεση στην ε, ε, ένταξη μεν, χωρίς όμως να υποκαθιστά και τον διάλογο για τις προταξιακές διαδικασίες κλπ. Και το διάλογος αυτός θα πρέπει να αρχίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις Αθηνών με Σκόπια, εδώ η άποψή του είναι ότι πρέπει να βρεθεί λύση πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Λέει ότι θα μπορούσαν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει πριν λυθεί το θέμα του ονόματο και το θέμα του ονόματο να λυθεί παράλληλα με τι ε, διαπραγματεύσει σε ένα αρχικό στάδιο των διαπραγματεύσεων αυτών. Το γεγονό ότι και δύο πλευρέ πρόσφατα είπαν ότι ίσως ένα μνημόνιο κατανόησης να μπορεί να υπογραφεί ε, καλών σχέσεων γυτνίασης, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένα θετικό βήμα και το βλέπει θετικά. Τώρα επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Α, θα μιλήσω εδώ τώρα εκ μέρους... Θα ήθελα επίσης να τονίσω το εξής. Είναι είναι δύσκολα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στην περίπτωση της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αλλά νομίζουμε ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπήρξε πάντα μια θετική αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Υπήρξε μια σειρά από προβλήματα τα οποία έχουμε αναφέρει στα, σε σχέση με τα θέματα αυτά μεταξύ Βουλγαρίας και πρώην Σλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και έχουμε επιλύσει κάποια από αυτά. Παραμένουν όμως κάποια θέματα σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζεται της μίας χώρας από την άλλη από τα μέσα ενημέρωσης. Και όλα αυτά οδηγούν σε δυσκολίες. Τα δικαιώματα των εθνοτικά Βουλγάρων στη Μακεδονία Είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην εθνοτική ομάδα των Βουλγάρων στην Μακεδονία και οι οποίοι, οι οποίοι υφίστανται πιέσεις. Κατά την ε, επίσης υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια καλύτερη παρακολούθηση όλων αυτών των προβλημάτων και να υπάρξει μια καλύτερη διαδικασία όχι μονάχα με την ε, Ελλάδα αλλά και με την Βουλγαρία σε σχέση με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν ξέρω αν εσείς κύριε Πρέσβη θα μπορούσατε να εξασφαλίσετε να υπάρξει μια προσέγγιση των δύο κυβερνήσεων και να υπάρξει κάποιος διάλογος, κάποια αρχή διαπραγματεύσεων μεταξύ Βουλγαρίας και πρώην Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε ένα επικοδομητικό διάλογο μέσα στον οποίο μπορούν να υπερπηδηθούν όλα αυτά τα προβλήματα και αυτό φυσικά να γίνει πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης. Αυτό θα ήταν λοιπόν μια καλή προϋπόθεση για να μην υπάρξει κάποια αρνητική στάση από την πλευρά της Βουλγαρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίγενιν, λέει και ο πρόεδρος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, λέει ο κύριος Πρέντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την παρουσίαση που έκανε. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να γίνει αρκετά δύσκολη. Όπως γνωρίζουμε και αναφέρθηκε, είναι ο τέταρτος χρόνος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις ίδιες προτάσεις για τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση είναι δύνατο όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια στο τέλος να μην γίνει τίποτα. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις, τι σημειώσαμε. Το διμερές, ε, διμερής συμφωνίας μεταξύ ΦΥΡΟΜ, το υπόμνημα συνεννόησης, μεταξύ, το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και ΦΥΡΟΜ, αλλά όπως είπε και ο Βούλγαρος συνάδελφος, υπάρχει και κάποια ένταση ακόμα που υφίσταται με τη Βουλγαρία, μεταξύ Φιρόμ και Βουλγαρίας. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα σαφέστατο. Θέλουμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με αυτή τη χώρα. Συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Επίτροπος ο κύριος Φούλε το ΦΥΡΟΜ χτυπά εδώ και χρόνια την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομόνωση αυτής της χώρας απλώς αυξάνει τον εξτρεμισμό. Τροφοδοτεί ουσιαστικά έναν άκρο συναισθηματικό διάλογο, φορτισμένο διάλογο μεταξύ ε, των Σκοπίων και των γειτόνων της χώρας. Αυτές είναι οι γενικές παρατηρήσεις που έχω. Εγώ τι κάνω, θέλω να ζητήσω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον πρέσβη όσον αφορά τις εκλογές που θα λάβουν χώρα ε, την άνοιξη του επομένου χρόνου. Όσον αφορά τον τύπο, μάλλον στον τύπο διάβασα, ότι πρέπει να, υπάρχει, να ασκείται πλήρω το δικαίωμα ψήφου. Υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε όμω ψηφοφόροι, ε, πολίτε μάλλον, που δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, διότι δεν έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα έντυπα ταυτότητα, τα βιομετρικά, τι βιομετρικέ ταυτότητε, τα ψηφ, ψηφιακέ ταυτότητε. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο. Θα ήθελα να ξέρω τι εξηγήσει δίδονται από τι τις αρχέ για αυτό το πρόβλημα. Πότε θα ζητεί Πρέπει να το θέσουμε επίσημα αυτό το ερώτημα, ίσως ε, αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές όμως. Το να μην δίνεται δυνατότητα σε κάποιους πολίτες να ψηφίσουν, θεωρώ ότι δεν είναι μια στάση, πώς να το πω, ισορροπημένη. Λοιπόν, θα, θα ήθελα κύριε Πρέσβη να το λάβετε αυτό υπόψη σας παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέντα. Ο κύριος Σωστάνη Μερίλης, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Κάποιες μικρές παρατηρήσεις που είναι πολύ σημαντικές από τη δική μου πλευρά. Οι εντάσεις μεταξύ Βουλγαρίας και πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αυτό δεν είναι καινοφανές φαινόμενο. αναφέρθηκε ο συνάδελφος στις ε, ε, τωρινές αυτές ε, εντάσεις, αλλά εδώ και 20 χρόνια υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια υπήρξε πάντα μία ε, στάση καλής θέλησης και αυτοσυγκράτησης από την πλευρά της Ιουκοσλαβίας έναντι της ε, Μακεδονίας. και είχαμε πάντα υποστηρίξει τις θέσεις της Μακεδονίας και το καλύτερο συμφέρον της χώρας αυτής. Αλλά οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ευδοκιμήσει. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι ορθό αυτό το οποίο λέγεται ότι η Μακεδονία αντιμετωπίζει θετικά τις σχέσεις καλές γειτονίες με τους γειτονές της. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν ισχύει. Πρόσφατα υπήρξε μια κοινή δήλωση του, Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και εκεί αναφέρεται ότι όλοι οι γείτονες της Μακεδονίας θα πρέπει ε, να εκφράσουν την ανησυχία τους για την πολιτική της Μακεδονίας στα θέματα γειτονίας. Οι Βούλγαροι στη Μακεδονία βρίσκονται σε μεγάλη πίεση, ενώ όλες οι άλλες εθνοτικές ομάδες έχουν πλήρη δικαιώματα. Οι Αλβανοί, οι Ρωμά, όλοι αυτοί δεν έχουν προβλήματα, αλλά οι Βούλγαροι βρίσκονται υπό πίεση, γιατί στην ε, Μακεδονία υπάρχει ένα πρόβλημα ταυτότητας, γιατί οι αρχές στην Μακεδονία εδώ και δεκαετίες έχουν ακολουθήσει μια πολιτική αποβουλγαροποίησης. Και τώρα βλέπουμε να λαμβάνει η χώρα μια περαιτέρω διαδικασία μια διαδικασία επαναβουλγαροποίησης, μια προσπάθεια επαναβουλγαροποίησης από μέρες. Όλα αυτά τα λέω γιατί εγώ θα ήθελα οι αρχές της ε, Μακεδονίας να καταβάλουν όλες τις προσπάθειες οι οποίες περνάνε από τα χέρια τους ώστε να τροποποιηθεί και το σύνταγμα της χώρας αυτής το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των εθνοτικών ομάδων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να είναι το κράτος αυτό είτε ένα κράτος μόνο αυτών που έχουν μακεδονική ταυτότητα κατά την άποψή τους ή ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να δέχεται την πολυμορφία όλων των πολιτών που ζουν στη χώρα αυτή ανεξάρτητα από την εθνική της προέλευση. Αλλιώς είναι διακριτικού χαρακτήρα αυτό το σύνταγμα. Δεν θέλω τώρα να σταθώ στη δυνατότητα βέτο από την πλευρά της Βουλγαρίας αλλά η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρωμανία έχουν καθίσει μια πάρα πολύ σοβαρή θέση για τα θέματα αυτά, λέγοντας ότι οι πολιτικές ελίτ στην Μακεδονία φαίνεται αυτή τη στιγμή να ακολουθούν μια πολύ λανθασμένη και μη σόφρονα πολιτική. Εμείς θα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Τι θέλουμε τώρα, θέλουμε να έχουμε την ενταξιακή προοπτική να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ή προηγουμένως να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία αναφέρουμε σήμερα και μόνο μετά να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξη. Ούτω ή άλλως όμως τα προβλήματα αυτά θα αναδυθούν κατά τη διάρκεια τη διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ένταξη και θα αποτελέσουν βάρο και για την κυβέρνηση Μακεδονία. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Οπότε παρακαλώ κύριε Πρέσβη Όραφ να απαντήσετε στις παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τρία σχόλια ε, άκουσα και θα απαντήσω σε αυτά. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα. Ναι, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Συγχρόνω, αυτός ο διάλογος υψηλού επίπεδου βοηθάει η κοινωνία των πολιτών να βρεθεί πιο κοντά στην κυβέρνηση και να έχει την δυνατότητα να αναμειχθεί περισσότερο στις συζητήσεις. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Αλλά θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ κοντά το τι θα γίνει στη συνέχεια και θα Θέλαμε και εμείς να έχει περισσότερα δικαιώματα κοινωνία των πολιτών. Δεύτερον, τα προβλήματα με το διαβατήριο, το βιομετρικό. Μέχρι τώρα το πρόβλημα ήταν οι κατάλογοι, οι εκλογικοί κατάλογοι και οι ψηφοφόροι. Ποιος ήταν ο αριθμός των ψηφοφόρων. Ε, προσπαθήσαμε αυτό να το λύσουμε και μέσω του Οργανισμού για την ε, Ασφάλεια στην Ευρώπη. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και εμεί στην Αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα το παρακολουθήσουμε και αυτό παρετέρω. Τώρα, οι σχέσει καλή γειτονία με τη Βουλγαρία. Έχετε δίκιο. Χάθηκε πολλή χρόνο. Πολλά προβλήματα υπάρχουν και πρέπει να λυθούν. Και γι' αυτό ακριβώς τον διάλογο αυτό υψηλού επίπεδου προσχώρησης στην ε, συνάντηση που είχε η κυβέρνηση με την Κομισιόν συζήτησε και αυτά τα θέματα. Έγιναν δηλαδή κάποια βήματα. Ο Πρωθυπουργό Ποβό και έστειλε επιστολή στον ομολογό του και πρότεινε διάφορα βήματα. Βέβαια μπορεί κανείς να πει ότι αυτά δεν φτάνουν. Είναι όμως ένα βήμα. Κάτι έχει γίνει. Όπως είπατε, τα προβλήματα αυτά έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 20 χρόνια. Ελπίζουμε ότι εφόσον υπάρχει η βούληση, τα προβλήματα αυτά θα λυθούν τώρα σε λιγότερο από 20 χρόνια. Και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εγώ διαπιστώνω ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει τη βούληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Οπότε ολοκληρώνεται έτσι αυτό το σημείο, αλλά να σας ενημερώσω προηγουμένως ότι η Επιτροπή μας αφέρει θα έχει ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Χιρόμ, τον κύριο Ποπόφσκι, στις 27 Νοεμβρίου. Και μετά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο, κάθε επιτυχία στο απαιτητικό σας έργο. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 6 που είναι η ένταξη των μεταναστών και πώς επηρεάζεται η αγορά εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα που είναι ο εισηγητής για εισαγωγικά σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται περί γνωμοδότησης. Όσον αφορά την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, η συνάδελφος Χέρς της παρουσίασε το κείμενο. Κάπως ξεγελά ο τίτλος του κειμένου γιατί λέει ένταξη των μεταναστών και συνέπειες για την αγορά κλπ. κλπ προστίθεται ο συντονισμό όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρος ο τίτλος. Η πρώτη παράγραφος του κειμένου υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Και μετά αναφέρει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στους γείτονές μας εξ Ανατολών και εκ Νότου. Είναι αρκετά γνωστό αυτό. Ξέρετε ότι δημιουργούνται με αυτές οι σχέσεις με ομό και κύκλο και η γειτονία. Η γειτονία έχει πολύ σημαντικό λόγο, άρα και μας μας ε, συμφέρει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Πολύ μάλλον, πολύ μάλλον δε, διότι πολλοί από τους μετανάστες που καταφθάνουν στην Ευρώπη προέρχονται από εκεί. Δεν μπορώ να δεχτώ τις τροπολογίες που θέλουν να εξαλείψουν αυτές τις αναφορές. Δέχτηκα την παράγραφο, στη παράγραφο 2 μια μεταβατική φάση και τη δυνατότητα να δημιουργηθεί κοινή ατζέντα για την κινητικότητα, κοινό πρόγραμμα για την κινητικότητα και τη μετανάστευση. τρίτη παράγραφο, στην τρίτη παράγραφο συστήνω να μπαίνει μια η τυπική ρήτρα όσον αφορά συμφωνία σύνδεση για την κοινωνική ασφάλιση. Διότι υπάρχουν συμφωνίες όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση με κάποιες χώρες χωρίς να επηρεάζονται οι συμφωνίες σύνδεση. Έχω δεχθεί κάποιες σχετικές τροπολογίες, κυρίως του συναδέλφων Νικολάη, Βέμπερ και Λαμπέρ. Θα ήθελα μετά να υπογραμμίσω και κάτι άλλο να βάλουμε μια άλλη παράγραφο που ενθαρρύνει την Ένωση ούτως ώστε σε συνολικό επίπεδο να διοργανώνει συζήτηση επί του θέματος, συζητήσεις. Θα πρέπει να συζητηθεί ενδελεχώς, θα πρέπει να το συζητήσουμε και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Παράγραφος 4 λέει ότι εάν γίνεται σωστή διαχείριση της μετανάστευσης, με την κατάλληλη διαχείριση μετανάστευση, ιδίως η κυκλική μετανάστευση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων με τρίτες χώρες ε, ενισχύοντας την ε, καλύτερη βέβαια κατανόηση μεταξύ των επαφών μεταξύ λαών. Συνάδελφος Βέμπερ έκανε πρόταση μια τροπολογία που τη δέχομαι. Όμως την τροπολογία Παλέτσκης ε, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Είναι πιο δύσκολο να τη δεχτώ. θα προτιμούσα να μιλήσω για την παρέμβαση. Ε, όσον αφορά τις χώρες που είναι πηγή ε, ε, των μεταναστών, παρά να παρεύουμε άλλα μέτρα. Και νομίζω ότι η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών ετοιμάζει σχετικά μια γνωμοδότηση. Αυτά όσον αφορά την εξωτερική διάσταση του προβλήματος. Μετά υπάρχει μια άλλη τροπολογία η οποία αναφέρεται στα ωφέλη που έχει, θα μπορούσε να έχει αυτή η κυκλική μετανάστευση όσον αφορά τις μεταπολεμικές καταστάσεις. Ο πρώτος συμβιβασμός που παρουσιάζω ε, αφορά την παράγραφο 5 προτείνει να αυξήσουμε, να δεχτούμε που συναθίζουν 13, 14 και 15 να δεχτούμε μαζί αυτές και να τις ενώσουμε και να παρουσιάσουμε ένα κείμενο που επιτρέπει μια διεθνή προστασία για όποιον ζητά άσυλο. Μετά, η κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών της, εξω... της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και εκείνων που εργάζονται στις αντιπροσωπείες για να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα της μετανάστευσης. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, ειδική κατάρτιση. Αυτή η πρόταση, και εδώ κλείνω, Κλείνω εδώ μάλλον, τα είπα όλα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που υπέβαλαν. Έχουμε ακόμα χρόνο πριν την ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ Υπάρχει δυνατότητα διαλόγου προφανώς με διάφορους συναδέλφους. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ... Α, μάλλον ε, μπορώ να συζητήσω μαζί σας και τα θέματα υπάρχουν για την πρώτη παράγραφο. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Ευχαριστώ, κύριε Να δώσω το λόγο τώρα στους κύριους εισηγητές. Δεν μπορώ να το κάνω όμως αυτό γιατί δεν βλέπω πολλούς κύριους εισηγητές. Κλείνουμε έτσι τη συζήτηση αυτού του θέματος. Δεν σας κρατώ το λόγο γιατί δεν έχει νόημα. Με συγχωρείτε, κυρία Γκόμες. Κυρία Γκόμες. Ναι, απλώς θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου τον κύριο Πρέντα για την έκθεση που προετοίμασε. θα δω τις τροπολογίες και θα του δώσω τις ε, αντιδράσεις μου σε σχέση με κάποιες τροπολογίες οι οποίες μου φαίνονται κάπως ε, να μην συνάδουν με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μου. Μια από αυτές προέρχεται από ένα συνάδελφο της δικής μου ομάδας και λέει αυτή η τροπολογία Α, την έχει αποσύρει η τροπολογία. Ναι, συγγνώμη, τώρα το είδα αυτό. Στη χώρα μου, αυτοί οι οποίοι έχουν εργαστεί εκεί ως παράνομοι μετανάστες, έχουν υποστηρίξει την κοινωνική μας, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, διότι όντας παράνομοι παρόλα αυτά έδιναν τις εισφορές τους στην κοινωνική ασφάλιση. Το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι να ενισχύσουμε την ε, ε, διατύπωση στο κείμενο αυτό λέγοντας για τη συνεργασία με τις χώρες αυτές από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, να τους βοηθήσουμε να έχουν ένα σύστημα πραγματικής ε, νομικής προστασίας για τους ε, μετανάστες, παραγωγικά χώρες όπως η Λιβύη που είναι χώρες διέλευσης των μεταναστών, όπου υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να υποστηριχθούν οι χώρες αυτές για να μπορούν να, έχουν, να απολαμβάνουν ενός νομικού καθεστώτος και να προστατεύονται. Και επίσης φυσικά θα πρέπει να υπάρξει αυτή η διάκριση μεταξύ μεταναστών και προσφύγων. Θα ήθελα λοιπόν ο κ. Πρέντα να ενισχύσει λίγο περισσότερο την ε, διατύπωση που έχει χρησιμοποιήσει για τη συνεργασία με την ανώτατη αρμοστία για τους πρόσφυγες, ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η Σύμβαση των Ηνωμένων <clears throat> για τους πρόσφυγες. Όλα αυτά δεν είναι μονάχα θέμα ενθάρρυνσης, θα πρέπει να είναι προϋπόθεση, ώστε όχι μονάχα οι δικοί μας λαοί αλλά και οι εταίροι λαοί να το λαμβάνουν αυτό στην υπόψη σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν λίγο πρόωρο αυτό που σας είπα. Η συζήτηση πράγματι αρχίζει να ζεσταίνεται. Και θα δώσω λόγο στην κυρία Μουνίθ Ουρκίσα. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις εισηγητές συμμερίζονται απόλυτα τις απόψεις της συντονίστριας από την σοσιαλιστική ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως τον κύριο Πρέντα για την παρουσίασή του. Όλα αυτά είναι πολύ επικοδομητικά, πολύ ενδιαφέροντα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι πολύ επικοδομητική η στάση του τώρα για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Υπάρχουν δύο βασικές ιδέες. Το ένα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα ε, βρίσκονται σε κρεμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ασφάλιση απέναντι σε τρίτες χώρες. Επίτα, η ομάδα μας θεωρεί θετική την πρόταση να συμπεριληφθεί μια τυποποιημένη ρήτρα για το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, τις διάφορες συμφωνίες σύνδεσης με τρίτες χώρες που βασίζεται σε ίση μεταχείριση, ε, συντάξεις κλπ. Τώρα για τη γνωμοδότηση. Συμφωνούμε γενικά με την πρόταση του κυρίου Πρέντε και θα υπερψηφίσουμε τις δύο συμβαστικές τροπολογίες. Πιστεύουμε ότι όντω συμπεριλαμβάνουν πάρα πολύ καλά ε, διάφορες τροπολογίες που είχαν υποβληθεί στα δύο άρθρα τα πιο επίμαχα αλλά και που είναι τα πιο ουσιώδη του κειμένου. Όπω έχουμε πει και στον εισηγητή, θα ζητήσουμε για δύο παραγράφου την ψηφοφορία, την παράγραφο 1 και την παράγραφο 6. Στην παράγραφο 1 δεν πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αναφερόμαστε ε, στο more for more, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι πλήττεται περισσότερο πληθυσμός ο οποίο υποβάλλεται σε κινητικότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρε οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει την κινητικότητα του πληθυσμού αυτού να την εξαρτήσουμε από τις πρόοδους που κάνουν οι χώρες. Αντί να αρνηθούμε δηλαδή τον διάλογο που θα επιτρέψει στους πολίτες των χωρών αυτών να αντιμετωπίζονται επίσης όρες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Να προωθήσουμε το διάλογο ώστε να επωφεληθούν οι πολίτες αυτοί από τις αρχέ τις οποίε εμεί πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι είναι οι αναγκαίε για ολόκληρο τον κόσμο. Στην παράγραφο 6 τώρα. Πέρα από το να ζητάμε από τις χώρες προέλευσης να στηρίξουν του επίδοξου μετανάστε με την παροχή πληροφοριών και την παροχή κινήτρων για κυκλική μετανάστευση, να πούμε να συνεργαστούν με το πόρταλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση. Πιστεύουμε ότι είναι καλό να ζητάμε από τρίτε χώρες να συνεργάζονται στο πόρταλ αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να δίνουν ε, και κίνητρα στους πολίτες τους προκειμένου να αποφύγεται διαρροή εγκεφάλων. Τέλος για την τροπολογία αριθμός 1. Πιστεύουμε ότι ναι, αναφέρουμε όλες ε, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατά προτεραιότητα χώρες, στρατηγική σημασία με τη Λατινική Αμερική για παράδειγμα που είναι στην πρόταση γνωμοδότησης, αλλά ή που θα τις αναφέρουμε όλες ή που δεν θα αναφέρουμε καμία γιατί υπάρχουν ε, και οι χώρες στα Σούρια, Αφρική, η στρατηγική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιφέρειες, περιοχές του κόσμου που παίρνουν μετανάστες ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι ή που δεν πρέπει να αναφέρουμε καμία περιοχή και καμία χώρα ή πρέπει να τις αναφέρουμε όλες. Κατά τα άλλα συμφωνούμε με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέντα, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Ναι, Πρόεδρε, θα πω λίγα λόγια για το θέμα. Χαίρομαι που απεσύρθη η τροπολογία 9 Παλέσκης. Μόλις τώρα το έμαθα, ευχαριστώ όμως. Όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Γκόμες, Ευχαριστώ για αυτά που μας είπε και θέλω να πω ότι όπως είχα πει και εγώ όταν μίλησα αρχικά στην αρχική μου παρέμβαση πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες μέχρι ότου διεξαχθεί ψηφοφορία πιστεύω ότι έχουμε ακόμα χρόνο για να βρούμε μια λύση αποδεκτή όσον αφορά τη διατύπωση της πρώτης παραγράφου. Συμφωνούμε. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε από αυτό τελικά. Κάνει μια πρόταση ο κύριος Βέμπερ όσον αφορά την τροπολογία 1. Μετά ακούσαμε και τις παρατηρήσεις της κυρίας Μουνίφ. Πιστεύω ότι ήταν σωστά αυτά που υπόθηκαν. Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια βολική διατύπωση ούτω ώστε να γίνεται αποδεκτή από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Οπότε τώρα περνάμε στο debriefing του κυρίου Βιγέννη, ο οποίος προείδευσε της αντιπροσωπείας στη Σερβία και το κοσυφοπέδιο της ΑΦΕΤ με τη ΣΕΝΤΕ. Πρώτα πήγανε στο Βελιγράδι, όπου συναντήθηκαν με τις αρχές, με την κοινωνία των πολιτών και με διεθνείς οργανισμούς και εκπροσώπους τους. Και στη συνέχεια στην Πρίστινα, όπου συναντήθηκαν και πάλι με τις τοπικές ε, αρχές και τους τοπικούς παράγοντες. Έχουμε βέβαια προηγουμένως την έκθεση πρόοδου για την ε, διεύρυνση. Πήγαν εκεί ακριβώς για να δούνε τι πρόοδος έχει επιτευχθεί και πώς πάει ο διάλογος ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα. Η εξομάλυνση της σχέσης αυτής είναι στοιχείο κλειδί για την συνέχιση της διαδικασίας ε, Ολοκληρωσή και για τις δύο αυτές πλευρές. Πρέπει να λυθούν διάφορα εσωτερικά θέματα προκειμένου να προετοιμάσουμε τις δικές μας εκθέσεις που υπέβαλαν αυτή τη βδομάδα οι δύο εισηγητές και θα συζητηθούν στην ΑΦΕΤ το Δεκέμβριο. Κύριε Βίγενεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας για την δικιά σας συνεισφορά στην προετοιμασία των επισκέψεων αυτών είχαμε συναντηθεί πιο πριν. Λίγες εβδομάδες δηλαδή πριν πάει, πριν πάει η αντιπροσωπεία για τα Δυτικά Βαλκάνια εκεί. Η στιγμή πάντως της επίσκεψης πιστεύω ότι ήταν πολύ κατάλληλη και γιατί ήταν ε, πριν από την έκθεση πρόοδου της Κομισιόν αλλά και ήταν 100 μέρες ε, μετά ε, αφού δηλαδή ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα η κυβέρνηση, υπήρξε νέα κυβέρνηση εκεί. Πήγαμε λοιπόν και στο Βελιγράδι και στην Πρίστινα. Εμείς πήγαμε βέβαια νωρίτερα για να, τα... είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι καλά προετοιμασμένα. Και σίγουρα το μήνυμα το οποίο περάσαμε στους ομολόγους μας ήταν προς την κατεύθυνση που θέλαμε. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες βέβαια γιατί υπάρχει γραπτή έκθεση και εκεί θα βρείτε διάφορες λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επίσκεψη προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά. Συναντηθήκαμε με όλους τους βασικούς ε, φορείς, με εξαίρεση τον κύριο Νικολιβίτς, ο οποίος έλειπε στο εξωτερικό και γι' αυτό και δεν συναντηθήκαμε μαζί του. Η γενική πάντως εντύπωση από την ε, συνάντηση αυτή στη Σερβία είναι ότι η κυβέρνηση σημερινή Παρά τις ανησυχίες μας, όταν δημιουργήθηκε πριν από 100 μέρες περίπου δηλαδή πριν, διαπιστώσαμε ότι είναι έτοιμη να φέρει αποτελέσματα, παίρνει στα σοβαρά τις δεσμεύσεις της και συνεχίζει τον ε, διάλογο στο υψηλό πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο. Αυτή είναι μια άλλη απόδειξη για το ότι προχωράει στις υποχρεώσεις της. Πολύ βασικό αυτό. Βέβαια είναι πιο εύκολο ο ρόλος τους γιατί το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι υπέρ της Ευρώπης. Άρα δεν θα αντιταθεί σε βήματα που θα αναλάβει η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί στις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει και το διάλογο ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο ένταξη της χώρας στην Ευρώπη είναι κύρια προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης. Είναι κάτι που το πιστεύουν όλοι οι ηγέτες και των τριών κυρίων κομμάτων που συμμετέχουν ε, στο συνασπισμό ο αναπληρωτής Βούτσιφ που είναι υπεύθυνο για την ευρωπαϊκή ένταξη ε, το τονίζει. Γι' αυτό έχουν φροντίσει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή, θα μπορούσαμε να πούμε, για να προχωρήσει αυτό. Σε διάφορες συναντήσεις που είχαμε διαπιστώσαμε την ετοιμότητα και των μελών της δίκησης σε διάφορα επίπεδα. Φαίνεται ότι και το κύριο κόμμα το συναψισμό που δεν ήταν πολύ ισχυρό για καιρό είναι έτοιμο, παρόλο που συνήθως οι καινούργοι χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στα νέα τους καθήκοντα. Όμως και αυτό το κόμμα και η αντιπολίτευση μέσα σε λίγο παραπάνω από τρεις μήνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε, ενώ στην αρχή ασχολήθηκαν με τα εσωτερικά τους προβλήματα, τώρα έχουν λυθεί φαίνεται αυτά. Και έτσι στα τέλη του μήνα το Δημοκρατικό Κόμμα θα έχει νέα ηγεσία και θα αρχίσει να δουλεύει ως επικοδομητική αντιπολίτευση στη Σερβία. Θα ήθελα να σας μιλήσω για μια συνάντηση που είχαμε και αυτή ήταν με τον ηγέτη του κόμματος, του κύριου κόμματος που είναι στην κυβέρνηση, τον κύριο Βούτσιτς, ο οποίος έδωσε την εντύπωση ότι είναι σοβαρός πολιτικός και ότι επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στα αποτελέσματα παρά στις δεσμεύσεις. Όχι τόσο στις ε, δημόσιες σχέσεις ή στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στα αποτελέσματα. Τον προσκαλέσαμε να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έρθει εδώ και να μας μιλήσει για τις ιδέες του, τις υποχρώσεις που έχει αναλάβει, τις προθέσεις του εντυπωσιαστήκαμε γιατί μας είπε ότι δεν θέλει να έρθει για ένα σοου στις Βρυξέλλες, θέλει να έρθει για να καταφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα δηλαδή περιμένει να έχει αποτελέσματα και μετά να έρθει εδώ να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά. Μια άλλη σημαντική συνάντηση που μπορεί να ενδιαφέρει εδώ τα μέλη της Επιτροπής μας είναι η συνάντηση που είχαμε ψάχνω το όνομα γιατί δεν το θυμάμαι. Με τον κύριο Βούτσεβιτς, ο οποίος είναι εισαγγελέα και μας ε, εξήγησε τα επιτεύγματα της υπηρεσίας του. Συζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα για την προστασία των μαρτύρων, για τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε θέματα λαθρεμπορίου. Είναι δύσκολα βέβαια και βέστητα ζητήματα αυτά. Για τους αγνοούμενους επίσης μιλήσαμε. Η υπηρεσία του δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια και είπε ότι στην αρχή δεν περίμενε να έχει τόση πολλή δουλειά ήλπιζε ότι θα ήταν πιο εύκολο και πιο σύντομες οι διαδικασίες για να καταλήξουν σε αποτελέσματα. Τελικά όμως είχαν πολλές περιπτώσεις να εξετάσουν, υπήρχε δίωξη πολλών ατόμων και όσο περνούσε ο καιρός όλο και περισσότερο αφοσιωνόταν στο να ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του. Δεν ήταν σε θέση να μας πει βέβαια πόσο καιρό ακόμα θα κρατήσει η υπηρεσία του αυτή. Όσον αφορά τώρα τη σταθερότητα της κυβέρνησης, που τίθεται με κάποιο ερωτηματικό τον τελευταίο καιρό, φαίνεται ότι υπάρχουν καλές ε, σχέσεις εργασίας μεταξύ των ηγετών των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Και αυτό γιατί οι κύριοι στόχοι είναι κοινοί στην κυβέρνηση. Οπότε η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, δεν κινδυνεύει ότι ερωτήσεις υπάρχουν, εννοείται να θα σας απαντήσω, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ε, αυτής εξ αρχής, αλλά θέλω να περάσω τώρα στον επόμενο σταθμό της επίσκεψής μας, που ήταν Βόρειο Κωσυφοπέδιο, Gate 1. Ε, εκεί ενημερωθήκαμε από τη Γιούλεξ πρώτα απ' όλα, από την αποστολή Γιούλεξ εκεί. Και μετά στο Νοβοσέλο, στο σταθμό εκεί κάναμε έναν σύντομο σταθμό, ενημερωθήκαμε για τον ρόλο τους, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ούτε θα θέλω να πω σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να σας πω ότι ο επικεφαλής Ε, μάλλον ότι αργότερα στην Πριστίνα συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της Γιούλεξ, ο οποίος είπε ότι ίσως θα ήταν καλύτερη λύση αν ο ρόλος της Eurolex άλλαζε και μπορούσε να αναλάβει και τις ευθύνες της ε, K4 στο μέλλον, ώστε όλη η δομή και η δουλειά να διευκολυνθεί. Γιατί από ό,τι μας είπε, η, χρωμοδότηση έρχεται, η χρωματοδότηση έρχεται λίγο πολύ από τις ίδιες πηγές, αλλά φαίνεται ότι το θέμα αυτό δεν είναι προς εξέταση γρήγορα. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι το κοσυφοπέδιο και οι αρχές του ενθαρρύνονται από έκθεση σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι υπάρχουν οι για να αρχίσει και το καθεστώς διευκόλυνσης θεωρήσεων Οπότε αυτό το θέλουν πολύ. Μάλιστα, συγκεκριμένα ο υπουργό για την Ευρωπαϊκή Ένταξη είπε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι όλο και πιο δύσκολο οι άλλες περιοχές ε, στην περιοχή που προετοιμάζονται για το ίδιο πράγμα έχουν λιγότερους δείχτες να καλύψουν. Είναι πιο εύκολη δουλειά για αυτούς, όχι για μας, αλλά παρόλα αυτά ε, προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι αν τα καταφέρουμε σημαίνει ότι πραγματικά είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Πάντως μια πιο αισιόδοξη άποψη από τις σερβικές αρχές ο Πρωθυπουργό του Κωσυφοπαιδίου μας είπε να μην είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που κυβερνήσεις στην Σερβία ε, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, κάνουν υποσχέσεις, αλλά μετά δεν φέρουν σε πέρα στις υποχρεώσεις τους. Πάντως είναι ενθαρρυντικό. Είπε ότι ξεκινά διάλογος, αν μη τι άλλο. Τώρα κάτι διαφορετικό που θέλω να σας αναφέρω είναι ότι η συμμετοχή των Σέρβων που ζουν στο Κωσυφοπαίδιο, τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο, είναι ένα βασικό στοιχείο για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών Σερβίας και Κωσυφοπαιδίου. Είδαμε τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της δηλαδή, έναν Σέρβο που εξήγησε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τώρα προτείνουν μια αύξηση της ποσόστοσης των μειονοτήτων στο, στο Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου, δύο μέλη και ήταν αφαιρετικός και όταν συνεδεθήκαμε σε Σερβία με τον Βούτσεβιτς είπε ότι ήταν διατεθειμένος να συναντηθεί και με τον ε, Αντιπρόεδρο Σερβικής Καταγωγής και να συζητήσουν θέματα συμμετοχής στην ε, ενεργό πολιτική ζωή και την κοινωνική ζωή στο Κωσυφοπαίδιο. Πάντως το Κωσυφοπαίδιο αποτελεί βέβαια ακόμα ένα ε, σημαντικό θέμα. Οι Σέρβοι πάντως στο νότιο Κωσυφοπαίδιο συμμετέχουν στα κοινά είναι μια κάπως θετική εξέλιξη, θα έπρεπε να επεκταθεί και στο βόρειο κοσυφοπέδιο. Θα ήταν ο φυσικός τρόπος να λυθεί το πρόβλημα αυτό, το πιο φυσιολογικό. Η πρόκληση όμως παραμένει, γιατί εξαιτία των δομών του Κοινοβουλίου, των δομών γενικότερα, οι υπουργοί του Κωσυφοπεδίου, από ό,τι μάθαμε, δεν μπορούν να πάνε στο βόρειο Κωσυφοπέδιο, ακόμα και αν προσπαθούν να έχουν κάποια επαφή με τον κόσμο εκεί. Και βέβαια το κοσυφοπαίδιο θα παραμείνει ένα από τα θέματα τα οποία θα προσέχουν. Θα, πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη προσοχή και θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλε τι προσπάθειε για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε σχέσεις θετικές και διάλογο με τέτοιο τρόπο ώστε το Βόρειο Κόσοβο να είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού στερεώματος του πεδίου. Και ίσως θα έπρεπε να σταματήσω εδώ. Όπως σας είπα ήταν μια πολύ επίκαιρη επίσκεψη, πολύ θετική επίσκεψη και νομίζω ότι έχουμε πολύ θετικές εκτιμήσεις οι οποίες μπόρεσαν να γίνουν σε σχέση με τα τεκτενόμενα στο Κωσφοπέδιο και συγχρόνως στείλαμε και συγκεκριμένα και σαφή μηνύματα στους συνομιλητές μας τονίζοντας ότι τώρα πια ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ανοιχτός για τη Σερβία αλλά και για το Κωσφοπέδιο μέσα από την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αυτό σημαίνει ότι εφ' είναι στα χέρια των αρχών της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου να επιτύχουν τα απαιτούμενα και να δημιουργήσουν τις θετικές εξελίξεις οι οποίες θα δημιουργήσουν έφορο έδαφος για περαιτέρω πρόοδος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βηγενίν. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που ήταν μέλη της αντιπροσωπείας. Πρώτα ο κύριος Νταφ από την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Βίγενιν για τον τρόπο με τον οποίο προείδρευσε αυτή την αντιπροσωπεία. Όπως είπε, λειτουργήσε πολύ καλά, είχαμε μια καλή αντιμετώπιση. Και υπήρξε και πολύ καλή υποστήριξη από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και φυσικά και από τους ε, οι οικοδεσπότες μας και στο Βελιγράδι και στην Πριστίνα. Η δική μου εντύπωση που απεκόμισα είναι ότι στο Βελιγράδι κανείς πια δεν υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα είδος σιωπής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που δυνητικά μπορεί να είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη. Υπάρχει ένα κενό σε σχέση με την Ευρώπη και κάποιος θα πρέπει να καλύψει αυτό το κενό αν η πολιτική της Σερβίας πρόκειται να στραφεί με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ όμως με τον κύριο Βίγενιν όταν είπε ότι η νέα σερβική κυβέρνηση όσο παράδοξο και να φαίνεται είναι ικανότερη για να επιτύχει πρόοδο σε σχέση με το κοσυφοπαίδιο από ότι η προκάτοχος κυβέρνηση. Είναι σε πολύ καλύτερη θέση εσωτερικά, γιατί ξεκινά από μια πιο εθνικιστική θέση η οποία είναι ήδη γνωστή. Εάν λοιπόν θέλει να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις και στις παραχωρήσεις που ο κύριος Τάντιτς δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να κάνει, τότε θα έχουμε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη σε σχέση με το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά θεωρητικά, αλλά στην πράξη ήταν πολύ δύσκολο να ελοπιθεί. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υποτιμά κανείς τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στα σύνορα, στη διαχωριστική γραμμή. Όπως θέλετε να το λέμε αυτό το σημείο. Χρειάζεται να πετάνε με αεροπλάνο ή με ελικόπτερο τους ε, αστυνομικούς του Κωσυφοπεδίου στα σύνορα, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να διασχίσουν το βόρειο Κωσυφοπεδίο να πάνε στα σύνορα. και η Ulex η οποία έχει απεισχναστεί, έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού της, πρέπει να προστατεύεται από την K4 και αυτό κοστίζει περισσότερο για όλους μας. Το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του για την ULEX επισημαίνει ορισμένα ανησυχητικά σημεία που θα πρέπει να ερευνηθούν περισσότερο από εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πηγές ανησυχίας. Πιστεύω όμως ότι το πνεύμα της Ιουλέξ και η αποφασιστικότητά της να εκτελέσει το εγχείρημα για το οποίο βρίσκεται εκεί είναι αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο. Αυτό το οποίο αποτελεί θετική είδηση είναι ότι είναι, πιο εύκολο τώρα. Υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα επαφής μεταξύ των Σέρβων και των Κωσοβάρων Σέρβων. Υπάρχει μια καλύτερη λοιπόν δυνατότητα να υπάρξει μια γεφύρωση των διαφορών των δύο πλευρών και η συνέντευξη του κ. Βούτσιτς με τον κ. Πέτροβιτς ήταν πολύ θετική και πρέπει να διατηρηθεί αυτό το θετικό κλίμα δεν επαρκεί ο κύριος Ντούτσιτς να συναντήσει τον ομολογό του, θα πρέπει να υπάρξει και επαφή μεταξύ των Σέρβων και των Σέρβων του Κωσικοπεδίου. Γενικά, στο Κωσικοπεδίο αποκομίζει κανείς την εντύπωση ότι ακόμα δεν έχει καταδείξει η χώρα αυτή την ικανότητα να είναι μια χώρα αυτάρκης σε διοικητικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί στο παρελθόν δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο, να έχει, μια, να έχει τέτοιες δομές. Ήταν πάντα υπό τον έλεγχο κάποιου άλλου για τα τελευταία 500 χρόνια. Και η οι μεταρρυθμίσεις και ιδίως οι εκλογικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται πριν από τις εκλογές για το φθινόπωρο που θα λάβουν χώρα το φθινόπωρο του χρόνου θα είναι καλόδεχτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάφο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. συντομία πιστεύω ότι ήταν χρησιμότατη η επίσκεψη και μπορεί από αυτή την επίσκεψη να δούμε ότι χρειαζόμαστε και διάλογο και μεταρρυθμίσεις. Διτό στόχο. Αυτό είναι κάτι που απορρέει μάλλον από την επισκέψη. ενδεχόμενη εξομάλυνση σχέσεων Βελιγραδίου και Πρίστινας στα πλαίσια πλησιάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα που είναι σε τρία επίπεδα. Και αυτό είναι και αρμοδιότητα της, ε, εθνικ... της διεθνούς κοινότητας. Δεν είναι μόνο θέμα Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Ε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε πλέον την κυριαρχία και την ανεξαρτησία μέσω θεσμικής ε, παγίωσης και αποκέντρωσης. Μετά έχουμε δεύτερο επίπεδο που θα πρέπει να τεθεί σε διεθνή διάσταση. Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας η οποία θα πρέπει να αποφύγει τα διλήμματα της αναδιάθρωσης. σύμφωνα με τη 1244 το ΙΕ την απόφαση που δεν έχει εφαρμοστεί είναι πλέον εικονική. Ούτε και στο βόρειο κοσυφοπέδιο δεν εφαρμόζεται. Τρίτο επίπεδο. Πιο προβληματικό επίπεδο. Έλλειψη αναγνώρισης αυτού του σχήματος από πλευράς της σερβικής βορειοκοινότητας. 40.000 άτομα ζουν στη Βόρεια Μητρόβιτσα και σε διάφορες, ε, σε διάφορους δήμους. Και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσουν όθηση, ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα αυτά τα τρία επίπεδα. Μόνος τρόπος γι' αυτό είναι όπως έλεγα στην αρχή. Να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει το Κωσυφοπαίδιο και όχι μόνο αλλά και η Σερβία από αυτά που είδαμε και χρειάζεται συνεχής διάλογος. Σχέσεις Βελιγραδίου και Πρίστινας είναι κάτι στέρεο. Κυρίως διότι το, Βελιγράδιο, το Βελιγράδι θεωρεί δεδομένη την ευρωπαϊκή πορεία. Και αυτό θα είναι ευνοϊκό για τις σχέσεις των δύο χωρών, αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ. Και τέλος, η Ούλρικε Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Έντβαρτ Κούκαν. Ταυτίζομαι με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Και ευχαριστώ τον Κρίστιαν Βικένιν. Ήταν άριστος επικεφαλής αντιπροσωπείας και στις δύο χώρες. Αυτό το ταξίδι πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό για το έργο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, διότι επισκεπτόμενοι τις δύο χώρες στο χρονικό διάστημα μεταξύ της Χρυσομπορικής Επιτροπής, Επιτροπής για τη Διεύρυνση και της δικής μας ε, εκθέσεως ε, κατέστησε αυτή την επίσκεψη πάρα πολύ σημαντική. Ήρθα αργά και δεν άκουσα αυτά που είπε αρχικά και ο Σβιγγένιν. Ίσως το είπε. Ήμασταν εκεί πριν, ετοιμάζαμε το έδαφος για την Χίλαρη Κλίντον και την κυρία Άστον. ετοιμάσαμε το έδαφος, ετοιμάσαμε τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, κυρίως η Κάθριν Άστον. Δουλειά που έκανε και πριν και θα συνεχίσει και στο μέλλον. Να προσθέσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία πάνω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Στη Σερβία εξεπλάγην ευχάριστα, όπως πολλοί από μας. Είδαμε μεγάλη προθυμία από πλευράς νέας κυβέρνησης να προχωρήσει στο διάλογο με το Κωσυφοπέδιο και ο κύριος Τάτσης είπε σε κάποιες από τις συναντήσεις που είχαμε, είπε ότι είμαι εθνικιστής μεν, αλλά αυτό μπορεί να με βοηθήσει να προχωρήσω και να πίσω τους δικούς μου να προχωρήσουμε. Πρέπει να γίνουν πράγματα ακόμα, αλλά ο κύριος Βούτσης ήταν σαφέστατος. Είπε ότι τελικά θα τα καταφέρουν. Οπότε, θετικά τα μηνύματα από τη Σερβία προχωρούν προς εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσυφοπέδιο. Και οι Σέρβοι κάνουν προσπάθεια εξομάλυνση των σχέσεων. Δύο πράγματα έχω να προσθέσω για τη συνάντηση με τον κύριο Βούτσοβιτς. Ο κύριος Βίκαριτς ήταν αναπληρωτής. Τι με εντυπωσίασε. Το ίδιο το κτίριο με εντυπωσίασε. Πώς οικοδομήθηκε και είχε και ένα τμήμα συγκεκριμένο για την προστασία των μαρτύρων. Μπορούσαν οι μάρτυρες να μιλήσουν χωρίς να τους βλέπει κανείς, η είσοδός τους να είναι και αυτοί κρυμμένη. Καλό παράδειγμα, ελπίζω να χρησιμοποιηθεί με το σωστό, το καλύτερο τρόπο για να προστατεύονται μάρτυρες. Από κίνδυνο, να προστατεύεται η ταυτότητά τους όταν αυτοί είναι πρόθυμοι να μιλήσουν. Κάποιος... Α, μάλλον άκουσαν τις επικρίσεις που εκφράσαμε. Ότι υπήρχε ένας μάρτυρας στην εικαζόμενη υπόθεση για το εμπόριο οργάνων που μίλησε δημόσια και υποστήριζε τον Βουκοβίτς. Αυτό το κατακρίναμε, διότι έτσι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ενός μάρτυρα. Είπαν ότι ο μάρτυρας ήθελε να μιλήσει δημόσια ανοιχτά, ο ίδιος. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, μας είπαν. Θεώρησε ότι αυτό δείχνει λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και εργάζονται. Και κάτι άλλο που έθεσα εγώ και ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κινηθεί. Δεν έχω καταλάβει πώς όμως θα έπρεπε να κινηθούμε. Γιώβαν Ντίβιακ, υπόθεση Γιώβαν κάποιος ο οποίος τελικά άλλαξε πλευρά και υποστήριξε τους Βοσνίους, στρατηγός Οι Σέρβοι ζήτησαν να συλληφθεί και συνελήφθη πέρσι στην Αυστρία. Παρόλο που το Εθνές Ποινικό Δικαστήριο τον είχε αθώσει. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Στην Αυστρία είναι, στο Σεράγεβο είναι. Ο κ. Βούτσεβιτς σαφέστατα είπε ότι πρέπει να συμμορφωθεί με το σερβικό δίκαιο. Και ό,τι λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν ισχύει εκεί, το ο σερβικός νόμος ισχύει και χρειαζόταν να μνημόνιο συνεννόησης με τη Βοσνία όπως και με την Κροατία. Και δεν είναι πρόβλημα το, της εισαγγελία στην ε, Βοσνία, αλλά των πολιτικών. που δεν εφαρμόζεται το μνημόνιο αυτό συνεννόησης γιατί ούτε θα μπορούσαν να αλλάξουν οι διαδικασίες. Θα ήθελα να του δώσω συνέχεια αυτού του θέματος και να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή και στην ομάδα εργασίας. Στο Κωσυφοπαίδιο, τα είπαν οι συνάδελφοι. Αυτό που ήθελα να συζητήσω με τον Πρωθυπουργό Σάτσι, ακούστηκαν οι εικασίες φήμες ότι ίσως ε, να γίνει ένα σχηματισμό κυβερνήσει ε, και ίσω να διεξαχθούν και πρόορε εκλογέ χωρί να αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ότι είναι σταθερή κυβέρνηση. Εμεί είπαμε ότι αν δεν γίνει εκλογική μεταρρύθμιση μετά τι τελευταίε εκλογέ που δεν ήταν δίκαιε και ελεύθερε και είδαμε ότι υπήρξαν και κάποιε λαθροχειρίε, χωρί αλλαγή οι νέε εκλογέ δεν θα μπορούσαν να τύχουν τη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. για το Ιούλεξ. Τότε πηγαίναμε από το βόρειο Κωσυφοπέδιο μέσω Μητροβίτσας προς Πριστίνα και εξεδόθη τότε η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Με προβλημάτισε η αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης για την έκθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν έχει αποτύχει η Γιούλεξ. Και το κοσυφοπαίδιο έχει χρεοκοπήσει, αν θέλετε, εντό αγωγικών. Σαν υπόθεση. Εγώ προσπάθησα αυτά να τα αντικρούσω, διότι ήταν σαφής η επίκριση του ελεκτικού συνεδρίου. Είπε ναι δεν είναι τόσο καλή κατάσταση οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά στο κοσυφοπαίδιο, αλλά υπογράμμισαν ιδιαίτερα και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών επ' αυτού. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο ενωμένη όσο θα έπρεπε να είναι. Και ότι 22 έχουν αναγνωρίσει και 5 όχι κάτι μέλη και ότι δεν ε, στέλναμε αρκετά, αρκετό προσωπικό για τη Γιούλεξ αλλά και με πολύ καλά προσόντα και δεν ήμασταν ε, πρόθυμοι να αποσπάσουμε όσους χρειαζόταν. Και αυτό μας απασχολεί και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θέλουν τη Γιούλεξ, θεωρούν ότι είναι μεγαλύτερη πολιτική φύσεω αποστολή και έχει παραταθεί και η θητεία της αλλά δεν δίνουν την αναγκαία υποστήριξη. Ένα μέρος λοιπόν του προβλήματος σχετίζεται και με εμά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να στείλουμε και θα σταματήσω εδώ ευχαριστώντας σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Ευχαριστώ όλους σας που εκπροσωπήσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο καλά σε αυτή τη σημαντική περίοδο εξελίξεων και στις δύο χώρες το εκτιμούμε. Προχωράμε τώρα. Επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, που είναι τα διάφορα. Αλλά δεν βλέπω διάφορα στα διάφορα. Οπότε χρόνος και τόπος στην επόμενη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση ΑΦΕΤ θα γίνει Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, 7.30 το βράδυ. Συζήτηση με τον πρόεδρο της ΑΙΤ, τον κύριο Μαρτέλη. Μετά η συνεδρίαση που θα ακολουθήσει θα γίνει 5η 9 το πρωί και θα ψηφίσουμε στην εν λόγω συνεδρίαση. Το ψήφισμα για την Αλβανία και οι δύο συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα συνεδριάσεις. Γεια σας.